Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σχεδόν έχουμε εξαντλήσει το ακαδημαϊκό τέταρτο. Οι ε, ακροάσεις επειδή μοιάζουμε σεμινάρια ή με εργαστήρια, δηλαδή έχουν κάποιο ακαδημαϊκό χαρακτήρα, σεβόμαστε αυτό το ακαδημαϊκό τέταρτο. Ωραία δικαιολογία δεν έδωσε για την καθυστέρησή μας. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο σεμινάριο. Θερμό καλωσόρισμα απευθύνω προς τους καλεσμένους μας. Όπως είπα, έχουμε το σεμινάριο, το εργαστήριο με θέμα τη μεταρρύθμιση των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα οποροκυπευτικά. Τα οποροκυπευτικά αποτελούν νευραλγικό κλάδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και πολλά χρόνια και μάλιστα στηρίζονται από την κοινή αγροτική πολιτική. Είναι σημαντικό, σημαντική συμβολή των απορροκυπευτικών στη διατροφή και στην ποιοτική διατροφή. Έχουμε και εμείς ε, αναθέσει έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας στον κύριο Μέλλον και από το 2007 ε, έχουμε την εφαρμογή της ΚΑΠ και θα δούμε τις επιρροές της και τις επιπτώσεις αυτής της εφαρμογής στα απορροκυπευτικά. Όπως σας είπα, ο κύριος Μέλο είναι ο εισηγητής αυτή την έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας της ε, Επιτροπής Γεωργίας. Στόχος ε, του εργαστηρίου μας είναι να ακούσουμε κάποιες συστάσεις ε, για τη βελτίωση των ενωσιακών κανόνων ε, στον τομέα των απορροκυπευτικών και θα στηριχθούμε στην ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης που είναι αρκετά δυναμική εξελίσσεται Οπότε θα πρέπει να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των παραγωγών, των γεωργών και γενικώ του κλάδου. Θα ήθελα να καλωσορίσω τους καλεσμένους μας, τον κύριο Γιος Μπέιμαν από το Πανεπιστήμιο Wageningen των Κατοχωρών. Θα μας κάνει την πρώτη παρουσίαση στο εργαστήριο αυτό. Ξέρουμε ότι ο τομέας αυτός είναι σημαντικός στην Ολλανδία. Και η δεύτερη παρουσίαση θα γίνει από τους κυρίους Λουτσιάνο Τρεντίνη και Ζακ Ντάσκ από την Συνέλευση Ευρωπαϊκών Περιφερειών Παραγωγών Απορροκυπευτικών. Ο κύριος Μπέιμαν θα επικεντρωθεί κυρίως στα προβλήματα του κλάδου στις βόρειες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ οι δύο άλλοι καλεσμένοι μας θα επικεντρωθούν στην κατάσταση των απορροκυπευτικών στην Νότια κυρίως Ευρώπη. Ξέρετε ότι η ευρωπαϊκή γεωργία χαρακτηρίζεται από μεγάλη ποικιλομορφία. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη αυτές τις ε, ιδιαιτερότητες και τις διαφορές μεταξύ των χωρών. Γι' αυτό και διαιρέσαμε έτσι το εργαστήριό μας. Δεν ε, έχουμε δεν επιτρέπονται ομοιόμορφα μέτρα, μια και υπάρχουν τόσες ιδιαιτερότητε. Θα πρέπει να τις λάβουμε υπόψη. Αυτά. Εκ μέρου μου θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στον πρώτο μας καλεσμένο, τον κύριο Μπέιμαν. Αν είστε έτοιμος, περιμένουμε με ενδιαφέρον την παρουσίασή σας κύριε Μπέιμαν. Okay, thank you, Mr. Sikirski. Um, thank you for this. Uh... Ευχαριστώ πολύ για αυτή την, για αυτή την πρόσκληση. Ευχαριστώ τον κύριο Μασό, τον κύριο Ραγκόνο για την ε, διοργάνωση και για τη βοήθεια που μου έδωσαν προκειμένου να προετοιμαστώ. Είναι τιμή μου να σας παρουσιάσω ορισμένε από τις ε, ιδέες που κυκλοφορούν στις ε, βόρειο-ευρωπαϊκές χώρες σε ό,τι αφορά την ενδεχόμενη αναδιάρθρωση, τους ενδεχόμενους νέους κανόνες του καθεστώτος φρούτων και οπωροκυπευτικών. Έχω προετοιμάσει μια παρουσίαση, PowerPoint. Η παρουσίαση αυτή θα ξεκινήσει με τα βασικά συμπεράσματα Οπότε αν χάσετε τις ε, λεπτομέρειες αργότερα θα έχετε τουλάχιστον στο μυαλό σας από την αρχή τα συμπεράσματα. Δεύτερον, διαρθρωτικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα αυτή την εποχή στον τομέα σε όλη την Ευρώπη αλλά κυρίως στις ε, βόρειες χώρες. Τρίτον, θα δούμε κάποια στοιχεία για την ε, εξέλιξη του βαθμού οργάνωσης ε, η παραγωγή είναι οργανωμένη σε οργανώσεις παραγωγών, ε, τι μερίδιο διαθέτουν της ε, αγοράς στην Ευρώπη. Να υπογραμμίσω ότι εστιάζομαι κυρίως στις οργανώσεις παραγωγών διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο του κλάδου. και του καθεστώτος. Πρέπει να δούμε ποιες είναι αυτές οι οργανώσεις, πώς έχουν αναπτυχθεί, πώς εξελίσσονται, ε, πώς ε, επηρεάζουν, πώς έχουν επηρεάσει τα τελευταία δέκα χρόνια τον τομέα και πώς οι κανόνες του τομέα επηρεάζουν την, ε, ε, τις οργανώσεις παραγών. μετά θα προσδιορίσουμε κάποιες τάσεις σε ό,τι αφορά τις ε, γεωργικές, γεωργικούς συνεταιρισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν απαιτείται η ύπαρξη συνεταιρισμών από την ομοθέσια αλλά σε πολλές ε, χώρες αλλά σε πολλές χώρες έχει γίνει αντιληπτή η σημασία των συνεταιρισμών και στην εθνική τους νομοθεσία έχει προβλεφθεί η νομική μορφή του συνεταιρισμού, αλλά ακόμα και όταν δεν, έχουν, δεν έχει προβλεφθεί, οι συνεταιρισμοί υφίστανται στην πράξη. Πέμπτον, θα δούμε τις ε, εμπειρίες και ορισμένα προβλήματα του σημερινού καθεστώτος και τέλος θα καταλήξουμε σε συστάσεις. Καταρχήν να σας πω ποιος είμαι εγώ, να συστηθώ. Ε, είμαι επίκορος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Βάχενιγκεν. Είναι ένα σχετικά μικρό πανεπιστήμιο με 10.000 περίπου φοιτητέ. Αλλά είναι το αγροτικό και γεωργικό πανεπιστήμιο της, ε, των κάτω χωρών. Παλιότερα ονομαζόμασταν γεωργικό πανεπιστήμιο, τώρα ονομαζόμαστε πανεπιστήμιο των επιστημών της ζωής. Ε, έχω εμπειρία στη διοίκηση επιχειρήσεων Έχω μελετήσει το καθεστώς των φρούτων και των προεκπευτικών από την πλευρά των επιχειρήσεων. Θεωρώ ότι οι εκμεταλλεύσεις και οι οργανώσεις παραγωγών είναι επιχειρήσεις. Οπότε έχω συνδυάσει την οικονομία, τις πολιτικές επιστήμες και την θεωρία της οργάνωσης. Θεωρώ τον εαυτό μου εμπειρογνώμονα ειδικό στους, στους γεωργικούς συνεταιρισμού στην Ευρώπη. Πριν από δύο χρόνια ολοκληρώσαμε ένα project που ονομαζόταν στήριξη των γεωργών των ε, γεωργικών συνεταιρισμών ε, ήταν ένα project της ε, Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οκτώ διαφορετικές εκθέσεις επεξεργαστήκαμε για τους γεωργικούς συνεταιρισμούς σε όλη την Ευρώπη όλες αυτές οι εκθέσεις βρίσκονται στο, στη σελίδα του ίντερνετ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Πανεπιστημίου του Βάχενιγκεν. Ήταν πολύ ωραίο αυτό το project γιατί για πρώτη φορά στην ιστορία έγινε μια συνολική σφαιρική μελέτη των γεωργικών συνεταιρισμών σε όλη την Ευρώπη των 27. Αυτά για μένα τώρα, τα συμπεράσματά μου. Από όπου ξεκινάμε κιόλας. Και εκεί θα τελειώσουμε κιόλας. Πρώτον, παρατηρείται μια ταχεία διαρθρωτική αλλαγή στον κλάδο των προκυπευτικών στην Ευρώπη. Οι εκμεταλλεύσεις μεγαλώνουν, ε, η εξειδίκευση αυξάνεται και αυτό σημαίνει ότι ε, αλλάζουν και οι απαιτήσει ε, των εκμεταλλεύσεων σε ό,τι αφορά τη στήριξή του από τις, εθνικές, από τις ε, ευρωπαϊκές αρχές. Δεύτερον, ο βαθμός οργάνωσης των παραγωγών σε οργανώσεις παραγωγών έχει αυξηθεί γρήγορα τα τελευταία δύο χρόνια, τα τελευταία δέκα χρόνια. Τα στοιχεία δείχνουν ότι έχουμε όλο και περισσότερους ε, παραγωγούς, γεωργούς που ανήκουν σε τέτοιες ε, οργανώσεις και όλο και μεγαλύτερο μερίδιο αντιπροσωπεύεται από αυτές. Βέβαια, υπάρχουν αρκετά μεγάλες διαφορές στο βαθμό οργάνωσης ε, μεταξύ των διαφόρων χωρών και αυτό ενδεχομένως οφείλεται σε αλλαγές που υπάρχουν, ε, διαφορές που υπάρχουν στην ανάπτυξη των συνεταιρισμών. Επίσης, άλλο συμπέρασμα είναι ότι δεν χρειάζονται νέοι κανόνες, ενδεχομένως κάποιες προσαρμογές των υφιστάμενων κανόνων. οργανώσεις παραγωγών που είναι θελοντικής φύσεως ε, πρέπει να έχουν πάντοτε χρόνο να αναπτυχθούν και να οριμάσουν. Αυτό που χρειάζονται οι γεωργοί και οι οργανώσεις παραγωγών είναι νομική ασφάλεια. Να ξέρουν πώς θα είναι η κατάσταση πέντε χρόνια μετά. Γιατί οι παραγωγοί και οι οργανώσεις παραγωγών κάνουν μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμε επενδύσει, Οπότε για αυτούς είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γνωρίζουν από τώρα τι θα αποδώσει η επένδυσή τους, ποια θα είναι η κατάσταση και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αυτών των επενδύσεων αν πάρουν για παράδειγμα μια ενίσχυση σήμερα κλπ. Θέλουν να ξέρουν πώς θα χειριστούν αυτές τις ενισχύσεις και πώς θα κάνουν τις επενδύσεις τους για το μέλλον. Ωραία. Να σας δώσω μερικά αριθμητικά στοιχεία καταρχήν για την ε, σημασία του τομέα στις βόρειες χώρες. Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορείτε να διαβάσετε τα νούμερα αυτά στην οθόνη, αλλά τα έχετε στο κείμενο το οποίο σας έχουμε μοιράσει, σε χαρτί. Αν δείτε τις πέντε πρώτες χώρες, Βέλγιο, Γερμανία, κατοχώρες Πολωνία και Ηνωμένο Βασίλειο, αυτές είναι οι βασικές χώρες μεγαλύτερη παραγωγή ε, φυτών και απορροκυπευτικών στο, στο βορρά. Και ε, τα καρότα είναι πολύ σημαντικό προϊόν, κρεμμύδια, τομάτες, ε, αγκούρια και απλώς φρούτων ε, αχλάδια και μήλα. Είναι σημαντικές λοιπόν αυτές οι παραγωγές χώρες για όλη την Ευρώπη. Τώρα, τι συμβαίνει. Έχουμε γρήγορη μείωση του αριθμού των εκμεταλλεύσεων. Ε, εδώ δεν βλέπετε την Πολωνία γιατί είναι τόσο πολλές οι εκμεταλλεύσεις εκεί που δεν θα, έμπαινε, χωρούσαν στο γράφημα αυτό. Ε, πάντως και εκεί βλέπουμε την ίδια τάση όλοι, όλες αυτές οι χώρες ε, παρουσιάζουν μείωση των εκμεταλλεύσεων. Βλέπετε αυτή είναι η τελευταία πενταετία εδώ, 2005-2010. Ε, στο κάτω χώρες μείωση 15%, Βέλγιο μείωση 18%, ε, ε, στην Γερμανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο παρόμοιες μειώσεις σε ορισμένες ε, χώρες ε, το 1 τρίτο των εκμεταλλεύσεων έχουν εξαφανιστεί. Ε, η παραγωγή όμως δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα. Το οποίο σημαίνει ότι μειώνονται οι εκμεταλλεύσεις αλλά αυξάνεται η, ε, η επιφάνεια κάθε εκμετάλλευσης. Ε, κάτω χώρες, πάρτε αυτή την διαφάνεια ε, είναι στα Ολλανδικά οι τίτλοι, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό που βλέπετε είναι ότι ο, ο, ο αριστερός άξονας, ο αριστερός κατακόρυφος άξονας ε, ε είναι ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων στις κάτω από 600 μέχρι βλέπετε κάτω από 400 σε 13 χρόνια ενώ η μπλε γραμμή είναι η μέση επιφάνεια, η μέση έκταση επιφάνεια κάθε εκμετάλλευσης. Το συμπέρασμα είναι ότι η, το μέγεθος των εκμεταλλεύσεων αυξάνεται με ταχύτητα. Συγγνώμη, η μπλε γραμμή είναι η μέση ε, έκταση εκμετάλλευσης που έχει αυξηθεί από 2 σε 6 περίπου εκτάρια σε 13 χρόνια η μέση επιφάνεια κάθε εκμετάλλευσης. Οπότε βλέπετε πόσο γρήγορα μεγαλώνει η εκμετάλλευση και γίνονται πιο επαγγελματικέ. Τώρα, περνάω στο βαθμό οργάνωσης των γεωργών σε γεωργικές ε, οργανώσεις. Αυτά είναι στοιχεία της Κομισιόν από την έκθεσή του 2014. Δείχνει ότι υπάρχουν διαφορές στο βαθμό οργάνωσης στα διάφορα κράτη-μέλη. Ο μέσος όρος σε όλη την Ευρώπη είναι 43%. Μερικές χώρες έχουν πολύ ψηλότερο βαθμό οργάνωσης ενώ άλλες χώρες έχουν πολύ χαμηλότερο βαθμό οργάνωσης. Πώς το ερμηνεύουμε αυτό. Ενδεχομένως το σύστημα λειτουργεί καλύτερα σε κάποιες χώρες και χειρότερα σε κάποιες άλλες. Παρ' όλα αυτά θα ήμουν πολύ προσεκτικό σε σχέση με αυτό το συμπέρασμα και θα σας εξηγήσω γιατί σε λίγο. Αν δούμε τα, τα λεπτομερή ε, αριθμητικά στοιχεία, πιο συγκεκριμένα τις αναγνωρισμένες ε, οργανώσεις παραγωγών το μερίδιο των οπροκυπευτικών και, την αξία της παραγωγής ε, ίσως δεν, βλέπετε εύκολα αυτά τα νούμερα οπότε τα έχω βάλει σε ένα γράφημα η μπλε γραμμή εδώ είναι ο αριθμός των παραγωγών που είναι μέλη μιας αναγνωρισμένης οργάνωσης παραγωγών αυτό το ποσοστό αυξήθηκε από το 10% ως το περίπου 16% την περίοδο 2004-2010 σημαντική αύξηση, όχι βέβαια εξαιρετικά ψηλή, αλλά γιατί ξεκινήσαμε πολύ χαμηλά. Η σημαντική γραμμή μου είναι η κόκκινη. Η καμπύλη αυτή που είναι το μερίδιο ε, της συνολικής αξίας των προκυπευτικών ε, που πωλείται μέσω οργανώσεων παραγωγών. Ε, αυτό το μερίδιο που κατέχουν οι οργανώσεις παραγωγών στη συνολική αγορά οπωροκυπευτικών αυξήθηκε από 30 περίπου σε 44% από το 2004 στο 2012. Ε, είναι σημαντική αύξηση. Δεν έχει διπλασιαστεί βέβαια, αλλά έχει αυξηθεί και συνεχίζει να αυξάνεται. Οπότε, είναι προφανές ότι η, ε, το σύστημα, το καθεστώς των οπροκυπευτικών ε, οθεί τους γεωργούς να ενταχθούν σε οργανώσεις παραγωγών και να πολλούν τα προϊόντα τους στην παραγωγή τους μέσω των οργανώσεων αυτών. Τώρα, αυτό το γράφημα συγκρίνει το βαθμό οργάνωσης του 2004 με το βαθμό οργάνωσης του 2012. Το 2004 έχουμε δημοσιευμένα στοιχεία, το 2012 ε, δεν έχουμε δημοσιευμένα στοιχεία, τα πήρα από μια παρουσίαση εκπροσώπου της Κομισιόν. Οπότε δεν είναι επίσημα, αλλά φαντάζομαι ότι είναι σωστά για να τα παρουσιάζει η Κομισιόν δημόσια. Αυτά τα στοιχεία δείχνουν σαφώς ε, οι κόκκινες, οι κόκκινες είναι το 2004 και οι άλλες είναι το 2012. Ε, φαίνεται ότι ο βαθμός οργάνωσης έχει αυξηθεί σε όλες τις χώρες, εκτός ενδεχομένως από την Ελλάδα και ίσως και το Ηνωμένο Βασίλειο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο είχαμε προβλήματα με την αναγνώριση των οργάνωσεων παραγωγών. Με αυτές τις εξαιρέσεις όλες οι άλλες χώρες έχουν παρουσιάσει αύξηση του βαθμού οργάνωσης. Μάλιστα στην Πολωνία, Τσεχική Δημοκρατία, Ισπανία, Γερμανία, η Αυστρία, Ιταλία, έχουν ε, δώσει πολύ, μια πολύ μεγάλη αύξηση του βαθμού οργάνωσης. Οπότε φαίνεται ότι το σύστημα προκυπευτικών έχει πραγματικά πετύχει στο να οθήσει τους παραγωγούς να γίνονται μέλη των παραγών. Για τις κάτω χώρες, να δούμε το παράδειγμα, είχαμε πάντοτε ψηλό βαθμό οργάνωσης, ε, ξεκινήσαμε στο 65% περίπου το 2000, 2002 και φτάσαμε μέχρι το 90% το 2009. Ε, μετά μειώθηκε λίγο ο βαθμός οργάνωσης ε, και το ίδιο ενδεχομένως θα αναμένουμε και σε άλλες χώρες να συμβεί. Για ποιος είναι ο λόγος. Ε, ο λόγος της μείωσης του βαθμού οργάνωσης τα τελευταία χρόνια, 2010-2011, δεν έχουμε στοιχεία πιο αργά, ίσως θα μειωθεί ακόμα περισσότερο βέβαια. Ε, ο λόγος είναι ότι ορισμένες ε, εκμεταλλεύσεις γίνονται πια τόσο μεγάλες που δεν επιθυμούν να είναι μέλη οργανώσεων παραγωγών. Θεωρούν ότι είναι ανταγωνιστές των συναδέλφων τους πλέον και όχι πραγματικοί συνάδελφοι. Μιλάμε για εκμεταλλεύσεις 50 εκταρίων, ε, παραγωγή σε θερμοκήπια, Ενδεχομένω δεν χρειάζεται να είναι μέλη οργανώσεων παραγωγών, διότι είναι τόσο ισχυρέ πια αυτέ οι εκμεταλλεύσει που ε, μπορούν να τα βγάλουν πέρα ε, ανεξάρτητα από μόνες του. Οπότε σε ορισμένε βόρειε βορειοευρωπαϊκές χώρε αυτό θα συμβεί. Δεν θεωρώ ότι είναι αρνητικό φαινόμενο είναι ένα γεγονός απλώ οι εκμεταλλεύσει αυτές γίνονται τόσο μεγάλες που δεν χρειάζονται την συνδρομή των οργανώσεων παραγωγών για να εξασφαλίσουν μερίδε στην αγορά και θέσεις στην αγορά. Α προχωρήσουμε να δούμε τα στοιχεία που προέκυψαν από μια προηγούμενη μελέτη την οποία ανέφερα για, την, για τους συνεταιρισμούς. Όπως σας είπα, οι οργανώσεις παραγωγών είναι ένας τύπος συνεταιρισμού ε, μερικές φορές ταυτίζονται από νομικής πλευράς ε, με συνεταιρισμούς. Ε, είναι λοιπόν χρήσιμο να συγκρίνουμε ε, τη συγκρίνουμε με άλλου τύπου συνεταιρισμούς. Αυτά τα στοιχεία τα έχουν πάρει από την έκθεση μέσα του 2012. Βλέπουμε τις διαφορές της σχετικής σημασίας των συνεταιρισμών στην ε, εμπορία των προϊόντων. Ε, Φιλανδία, Ολλανδία, Δανία είναι οι χώρες στις οποίες έχουν απτυχθεί περισσότερο οι συνεταιρισμοί. Από την άλλη μεριά έχουμε την Ουγγαρία, την Ελλάδα, τη Σλοβακία, Λιθουανία, Ηνωμένο Βασίλειο. Τα στοιχεία του Ηνωμένου δεν είναι σωστά δυστυχώς και μετά έχουμε Ρουμανία, Βουλγοριά, σχεδόν δεν έχουμε καθόλου συνεταιρισμού. Ε, ο μέσος όρος ε, στην, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 40%. Μιλούμε για όλα τα γεωρικά προϊόντα μαζί, δεν μιλάμε μόνο για τον κλάδο των προκυπευτικών. Μιλάμε για ε, κρέας, ε, μιλάμε για αυγά, για γαλακτοκομικά κλπ. Τώρα, να σας πω δύο λόγια για το, τα πορίσματά μας όταν εξετάσαμε τους συνεταιρισμούς. Αυτά τα συμπεράσματα έχουν σχέση και με την εξέλιξη των οργανώσεων παραγών και με οποιασδήποτε αποφάσεις περί πολιτικής ε, θέλουμε να λάβουμε. Πρώτον, το μερίδιο αγορά των συνεταιρισμών αυξάνεται. Αυτό είναι μάλλον θετικό. Ειδικά για αυτούς που θεωρούν ότι οι συνεταιρισμοί είναι κάτι καλό για τη γεωργία, τα μηνύματα είναι θετικά. Δεν έχω όμως ακριβή στοιχεία. Δεύτερον, ε, υπάρχει ανάγκη βελτίωση της διαπραγματευτικής θέσης των γεωργών και των συνεταιρισμών. Αυτό όμως είναι κλασικό πρόβλημα ε, οι υπεραγωγοί πρέπει να ενισχύσουν τη θέση τους σε σχέση με, τους ε, μεγάλους, με τις μεγάλες αλυσίδες που αγοράζουν τα προϊόντα τους. Γι' αυτό το λόγο, αυτό είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους μεγαλώνουν, μεγενθύνονται οι συνεταιρισμοί. Μερικοί γεωργοί, μάλιστα, ε, παραπονέθηκαν ότι οι συνεταιρισμοί γίνονται μεγάλες εταιρείε. Και πράγματι αυτό είναι ένα δίλημα για να είναι προσιλωμένοι και, και να δείχνουν πίστη οι γεωργοί στις, ε, στους συνεταιρισμούς τους, ε, να συμμετέχουν και να νιώθουν κοντά στο συνεταιρισμό τους, ε, πρέπει οι συνεταιρισμοί να παραμείνουν μικροί. Γιατί όταν μεγαλώνουν πάρα πολλοί οι συνεταιρισμοί, δεν γνωρίζουν το ένας με τον άλλο, δεν έχουν προσωπική επαφή. Από την άλλη μεριά, οι συνεταιρισμοί αυτοί όπως και οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση θα πρέπει να μεγαλώσει, να μεγαλώσουν προκειμένου να βελτιώσουν τη διαπραγματευτική τους ε, θέση. Οπότε αυτό είναι ένα δίλημα για όλους τους παραγωγούς, για όλους τους συνεταιρισμούς. Και δεν υπάρχει λύση. Μετά, ε, περισσότερη προσοχή στην κατακόρυφη ολοκλήρωση της αλυσίδας. Ε, η αλυσίδα γίνεται όλο και πιο ολοκληρωμένη. Τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι οι ε, γραφειοκρατικές διαδικασίες μειώνονται, τα προϊόντα μεταφέρονται κατευθείαν από την εκμετάλλευση στη, στο σημείο πώλησης ο πλευρά υγιεινή των τροφίμων και ασφάλιση των τροφίμων ε, είναι σημαντικό να ε, μειώσουμε ε, τις διαδικασίες ε, από το ένα στάδιο στο άλλο από πλευράς ε, ε, συμφερόντων του καταναλωτή επίσης χρησιμεύουν αυτή η ολοκλήρωση, είναι ωφέλιμη και αυτό και συμβαίνει. Και αυτό επηρεάζει και το πώς συνδέονται συμβατικά οι διάφορα, τα διάφορα επίπεδα μεταξύ τους. Τώρα, η ποιότητα της ε, ηγεσία ε, στους συνεταιρισμούς ε, έχει, είναι κρίσιμη σημασία. Είτε πρόκειται για το Διοικητικό Συμβούλιο, είτε πρόκειται για επαγγελματίες managers, είναι πάρα πολύ σημαντική, σημαντικός ο ρόλος τους για την επιτυχία των συνεταιρισμών. Και επίσης αυτό που είδαμε είναι ότι ε, είναι σημαντική η ευελιξία της νομοθεσίας για τους συνεταιρισμούς. Είναι πολύ σημαντικό η νομοθεσία να μην είναι ε, πάρα πολύ ε, στάσιμη και πάρα πολύ αυστηρή στις απαιτήσεις της. Ε, οι συνεταιρισμοί χρειάζονται ένα περιθώριο ευελιξίας για να αναπτυχθούν. Κοιτάω το ρολόι μου, να προχωρήσω λίγο. Εδώ βλέπουμε το... Ε, εδώ έχουμε συνδυασμό δύο διαφανειών. Καταρχήν είχα αυτό το slide ε, που είναι το μερίδιο αγορά των συνεταιρισμών στα κράτη-μέλη και μετά είδα το βαθμό οργάνωσης των φρούτων και και είδα ότι ο βαθμός οργάνωσης ε, του κλάδου σε ό,τι αφορά την αξία των προϊόντων που πολλούνται από οργανώσεις παραγωγών είναι μεγαλύτερος από, τον, από το μέσο συνεταιρισμό. Και αυτό σημαίνει ότι η πολιτική έχει πετύχει. Αν έχουμε τόσο πολλούς γεωργούς ε, με τόσο πολύ μερίδιο παραγωγής που πωλείται μέσω οργανώσεων παραγωγών, ε, μεγαλύτερο από ό,τι αντιπροσωπεύουν οι συνεταιρισμοί, τότε αυτό σημαίνει ότι οι οργανώσεις παραγωγών έχουν ενισχυθεί και έχουν αποκτήσει σημασία. Όχι βέβαια με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις χώρες, άλλες χώρες ε, ε, έχουν πιο ισχυρές, ε, πιο, ισχυρό, πιο υψηλό βαθμό οργάνωση άλλες πιο χαμηλό, αλλά παντού είναι πετυχημένο το σχήμα. Ωραία. Δύο ακόμα πραγματάκια θέλω να σχολιάσω πριν τελειώσω. Πρώτον, η εμπειρία με το ισχύον καθεστώς εξετάζοντας ε, όλες τις εθνικές αξιολογήσεις που υπάρχουν επίσης στο site της ε, Κομισιόν. Επίσης συζητήσαμε με εκπροσώπους του κλάδου και ορισμένες εθνικές αρχές στο Βέλγιο, τις κατοχώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία, τη Γερμανία, τη Δανία και την Αυστρία. Αυτά τα τέσσερα σημεία είναι τα πιο σημαντικά. Και ποια είναι. Ε, κάθε φορά που μιλάμε με οποιονδήποτε για αυτό το σύστημα, για αυτό το καθιστώς, ε, αυτό που προκύπτει πρώτο-πρώτο είναι ότι φαίνεται να υπάρχει νομική αβεβαιότητα, νομική ανασφάλεια. Στο πνεύμα του κανονισμού καταρχήν, της νομοθεσίας, συγγνώμη, όταν είχε συζητηθεί στη Διαχειριστική Επιτροπή η νομοθεσία αυτή, ε, ανάμεσα στην Κομισιόν και στις Εθνικές Αρχές, οι Εθνικές Αρχές είχαν αποκτήσει σαφή ιδέα για το ποιο ήταν ο στόχος, ποιο ήταν το πνεύμα της νομοθεσίας. Αλλά μετά όταν ήρθε το ελεγκτικό συνέδριο, ο, συγγνώμη, οι ελεγκτές τη Κομισιόν, οι ελεγκτές της Κομισιόν ερμήνευσαν διαφορετικά τους κανόνες. Και όλοι διαμαρτύρονται γι' αυτό. Ε, ο κλάδος χρειάζεται περισσότερη σαφήνεια, περισσότερο συντονισμό μεταξύ νομοθετών και ελεγκτών. Μετά, η αυστηρή ερμηνεία των κανόνων εξωτερικής ανάθεσης, του outsourcing. Τι σημαίνει εδώ εξωτερική ανάθεση, ποιο κομμάτι των δραστηριοτήτων διαχείρισης του προϊόντος μπορεί μια οργάνωση παραγωγών να αναθέσει σε μια εξωτερική εταιρεία. Υπάρχουν κανόνες γι' αυτό. Και πρέπει να γνωρίσουμε ότι οι οργανώσεις παραγωγών είναι και αυτές οι επιχειρήσεις που εξελίσσονται και ενδεχομένω ε, μπορεί να αλλάζουν τη στρατηγική τους. Έχουν συμβατικές εταιρείε με άλλες εταιρείε της αλυσίδας των τροφίμων, της τροφιμικής αλυσίδας και όλα εξαρτώνται από το πώ βλέπουμε του οργανώσει παραγωγών και ποιε είναι οι βασικέ του δραστηριότητε. Υπάρχουν δύο τύποι οργανώσεων παραγωγών. Μία οργάνωση παραγωγών που ε, απλώ διαπραγματεύεται ε, και δεν διαχειρίζεται τα ίδια τα προϊόντα. Και υπάρχει και άλλο, και άλλος τύπος οργάνωση παραγωγών που είναι πιο πολύ συνεταιριστικής φύσης ε, που ε, διαχειρίζονται τα ίδια τα προϊόντα. Για τις δεύτερες ε, δεν τίθεται τόσο πολύ θέμα εξωτερικής ανάθεσης, όμως οι πρώτες που είναι πιο πολύ διαπραγματευτικές οργανώσεις, ε, αυτές ε, αναθέτουν σε άλλες εταιρείες το μεγαλύτερο κομμάτι της, του χειρισμού των, των προϊόντων. Ξέρω ότι υπάρχει η επιθυμία να ενθαρρυνθούν οι διασυνορικές οργανώσεις παραγωγών, οι διεθνικές οργανώσεις παραγωγών, αλλά αυτό δεν είναι εύκολο. Ε, αυτό που είδαμε στις μελέτες μας, και τελειώνω, είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να δημιουργηθούν τέτοιες διεθνικές διασυνορικές οργανώσεις παραγωγών. Τέλος, ε, τα περιβαλλοντικά μέτρα είναι επίση πάρα πολύ υπερβολικά λεπτομερή, χωρίς σαφές αποτέλεσμα. Κλείνω εδώ ε, με κάποιες από τις συστάσεις μου. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το σύστημα προώθησης των ανάγνωσων παραγωγών έχει αποδειχθεί πολύ αποτελεσματικό. Ε, δεν φαίνεται επίσης να υπάρχει ανάγκη για νέους κανόνες. Υπάρχει όμως ανάγκη για περισσότερη νομική ασφάλεια και ε, λεπτομερής οδηγίες για το τι επιτρέπεται και τι όχι υπάρχουν αιτήματα απλοποίησης, ε, για παράδειγμα των περιβαλλοντικών μέτρων και αν ε, κάτι πρέπει να αλλάξει, αυτό θα πρέπει να είναι ίσως ενδεχομένως περισσότερη στήριξη της καινοτομίας, της επιμόρφωσης, τεχνική και οργανωτική βοήθεια κλπ. με το ανθρώπινο κεφάλαιο. Και τέλος, χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες, χρειάζονται περισσότερες λεπτομέρειες για το τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται από τους κανόνες ανταγωνισμού σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο ε, και καθώς επίσης και τι επιτρέπεται για την, για την ε, ε, σχέσεις μεταξύ οργανώσεων παραγωγών και ομάδων παραγωγών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Μπέιμαν. Ο λόγος τώρα στους επόμενους δύο καλεσμένους μας για τις δικές τους παρουσιάσεις. ένα λεπτό να λάβουν θέση. Φαντάζομαι έχετε συνεννοηθεί μεταξύ σας για το ποιος θα μιλήσει πρώτος και παρακαλώ να είστε σχετικά σύντομοι. Χωρίς μικρόφωνο, δυστυχώς, ο μιλητής. Καλημέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση και ευχαριστώ και τους ε, οργανωτές που έδωσαν ε, την ευκαιρία για αυτή την πολύ σημαντική συζήτηση για τα απορροκυπευτικά ένα κλάδο που ενδιαφέρει ολόκληρη την Ευρώπη. Ονομάζομαι Τρεντίνη, είμαι πρόεδρος της ΑΡΕΦΛ που είναι η συνέλευση Ευρωπαϊκών Περιφερειών Παραγωγών Απορροκυπευτικών και Καλοπιστικών ε, Φυτών. Καλύπτουμε 22 περιφέρειες ε, και 24% της παραγωγής της ο απορροκυπευτικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ιταλία μάλιστα έχουμε μία δομή συγκεκριμένη για τα απορροκυπευτικά και πολλούς ε, ιδιώτες ε, παρόχους. Τώρα, περνάμε στην παρουσίαση. Σε ό,τι αφορά τη δομή θα κάνω μια ανάλυση του περιεχομένου, της ε, έκθεσης και κάποιες προτάσεις που θα τις αναπτύξουμε στη συνέχεια. Θα ήθελα καταρχήν να πω δύο λόγια για την κατάσταση του κλάδου απορροκυπευτικού στον κόσμο, μετά στην Ευρώπη, με τις 27 χώρες. Για τα απορροκυπευτικά, μετά θα μιλήσω για τις οργανώσεις παραγωγών και τις ενώσεις οργανώσεων παραγωγών, πολύ σημαντικό θέμα για τον τομέα των απορρικρευτικών, ιδιαίτερα στο Νότο. Οι γνωστές οργανώσεις παραγωγών ε, διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στο σύστημα αυτό. Η διατήρηση και η περαιτέρω ανάπτυξη του κανονισμού, ιδιαίτερα για την κοινή οργάνωση αγοράς, είναι σημαντικές, γιατί οι κανόνες που έχουμε δεν χρειάζονται αλλαγή, ρηξικέλευθη, απλώς μερικές βελτιώσεις, κυρίως για να ληφθούν υπόψη τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της παραγωγής. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και επενδύσεις. Έχουμε σημαντική πρόοδο στα προκυπευτικά. Θα πρέπει να ενισχύσουμε λοιπόν το ρόλο των οργανώσεων των παραγωγών, να βελτιώσουμε τα επιχειρησιακά προγράμματα να προσέξουμε τις κρίσεις στις αγορές, ένα ιδιαίτερο πρόβλημα που κλώνησε και τις οργανώσεις των παραγωγών. Έχουμε τα περιβαλλοντικά θέματα, την καινοτομία που επίσης ενδιαφέρει τα απορρικτευτικά, προώθηση, διαφάνεια της αγοράς και προάσπιση και προώθηση της ευρωπαϊκής παραγωγής. Η κοινή οργάνωση αγοράς ε, μπορεί να συμπληρωθεί με διάφορες πτυχές της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ. Θα προσπαθήσω να είμαι λακολικός για να αφήσω λίγο χρόνο ε, και στους ε, συναδέλφους για τη συζήτηση. Έχουμε στην Ευρώπη το 17% της παγκόσμιας παραγωγής απορροκυπευτικών και βλέπετε τις ε, ραγδαίες εξελίξεις που είχαμε στην ανάπτυξη της παραγωγής στις διάφορες χώρες από το χάρτη που σας δείχνω. Σίγουρα έχουμε πολύ έντονη, έντονο ανταγωνισμό από τις χώρες της Αφρικής κυρίως 14%, ε, Νότια Αμερική 16%. Βέβαια έχουμε κάποια σύγκληση των αγορών Γι' αυτό και είναι επίφοβος ο ανταγωνισμός των άλλων φρουτοπαραγωγών χωρών. Βλέπετε στο χάρτη την παραγωγή οποροκυπευτικών κυρίως ε, στη Μεσογειακή Λεκάνη. Έχουμε την Ισπανία και την Ιταλία που αντιπροσωπεύουν περίπου το ίμιση της παραγωγής. Η Ελλάδα με τη Γαλλία μαζί αντιπροσωπεύουν το 16% της ευρωπαϊκής παραγωγής και μαζί με τις... Ε, οι χώρες αυτές ουσιαστικά είναι παράγουν 120 εκατομμύρια τόνους, ε, σχεδόν 70% της ε, κοινοτικής παραγωγής και περίπου 25% για την Ευρωπαϊκή Ένωση τζίρο. Τώρα έχουμε τις εξελίξεις από το 2007 μέχρι το 2011 με την εφαρμογή της κοινή οργάνωσης αγοράς βλέπετε τα στοιχεία για τις 27 χώρες μέλη και την ε, σημαντική αύξηση που παρατηρείται στις εξαγωγές των απορροκυπευτικών σε σχέση με τις εισαγωγές. Και αυτό ισχύει κυρίως για τα λαχανικά, αλλά και στα φρούτα παρατηρούμε παρόμοιες τάσεις. Είναι ενδεικτικό ότι αυτό είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των προϊόντων που επιτρέπουν στην Ευρώπη όχι μόνο να εισάγουν, αλλά όχι μόνο να εισάγει, αλλά και να εξάγει μεγάλους όγκους τέτοιων προϊόντων. Και μάλιστα οι χώρες του Νότου πρωτοστατούν στην παγκόσμια παραγωγή απορροκυπευτικών με μεγάλες δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη. Αναλύουμε το πλαίσιο της παραγωγής και την αξία της παραγωγής των απορροκυπευτικών και τη συμμετοχή ε, των οργανώσεων παραγωγών καθώς και των οργανώσεων παραγωγών. Έχουμε στην ε, Ευρώπη 22 δισεκατομμύρια ευρώ στις 28 χώρες, ενώ η συνολική παραγωγή των νοτίων χωρών είναι το 71% της ε, συνολικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλο σημαντικό στοιχείο που το ανέφερε και ο προελίσσας είναι η συμμετοχή των οργανώσεων παραγωγών και των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών και η διαφορά μεταξύ της, ε, του βαθμού οργάνωσης ε, στο βορρά και στο νότο. 47 εκατομμύρια είναι η αξία στη, στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 10 εκατομμύρια η αξία για τις νότιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 21% δηλαδή. Οπότε οι διαστάσεις και το μέγεθος των οργανώσεων παραγωγών και των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών βλέπετε είναι πολύ μικρότερο στο νότο σε σχέση με το βορρά. Και αυτό οφείλεται στον κατακαιρματισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και σε προηγούμενα πολιτικά συστήματα. Και Εξού και η διαφορά. Έχουμε τώρα ε, σημαντικά στοιχεία για τις μελλοντικές εξελίξεις. Ε, με βάση τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βλέπουμε ποιες ήταν οι εξελίξεις ε, στις αναγνωρισμένες και διαπιστευμένες ενώσεις παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών. 1643 στην Ευρώπη οργανώσεις παραγωγών, 83% δηλαδή, σε σχέση με το την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι απαραίτητη η, οργάνωση των παραγωγών για να αντιμετωπίσουν την παγκόσμια αγορά. Γι' αυτό και υπάρχει μια αυξητική πορεία της, του αριθμού των οργανώσεων παραγωγών και των ενώσεων. Ένας μεγάλος αριθμός οργανώσεων παραγωγών προϋποθέτει τη σύσταση και ενώσεων αυτών των οργανώσεων και 71% αυτών των ενώσεων των οργανώσεων παραγωγών βρίσκονται στη Νότια Ευρώπη. Κάτι που δείχνει την ε, ανάγκη της οργάνωσης που βιώνουν και ήδη οι γεωργοί. Μάλιστα, στόχος ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν το 60% της ε, οργάνωσης των γεωργών στην Ευρώπη. Και πλησιάζουμε προς το στόχο αυτό, όπως φαίνεται από τα στοιχεία που έχουμε. Και μάλιστα βλέπουμε τον, τον αριθμό των οργανώσεων παραγωγών που αυξάνεται με σημαντικούς ρυθμούς. Και βλέπουμε ότι οι ομάδες παραγωγών είναι 344 ε, και μόνο 50, στη, στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μόνο 57 στην Νότια Ευρώπη, που σημαίνει ότι δεν έχει αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό οργάνωσης και αυτό χρειάζεται κυρίως για την εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο αφορά τον αριθμό των παραγωγών, 323.000, οργανώσεις παραγωγών ή ενός παραγωγών, ε, στην Νότια Ευρώπη, ενώ στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 367.850. Ουσιαστικά 40% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, πάνω από ένα τρίτο, γύρω στο 1 εκατομμύριο δηλαδή, βρίσκονται σε κάποια μορφή οργάνωσης. Είναι σημαντικό αυτό γιατί έχουμε και πολλούς νέους επιχειρηματίες, νέους γεωργούς που θα συμβάλλουν στη δυναμική ανάπτυξη του τομέα των απορροκυπευτικών. Γιατί πολύ συχνά στην Νότια Ευρώπη οι γεωργοί είναι στις ηλικίες. Χρειαζόμαστε νέο αίμα. Και μερικά στοιχεία χρήζουν κάποιες διόρθωσεις, γιατί δημιουργήθηκαν και κάποιες ολιγομελείς οργανώσεις παραγωγών. Και καλό θα ήταν με τον κανονισμό να ενισχύσουμε τις ενώσεις των οργανώσεων παραγωγών και να δώσουμε την ευκαιρία και στις νέες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εφαρμόσουν μια πολιτική που θα προσαρμόζεται προς την κοινοτική και να ενταχθούν πολύ πιο γρήγορα στο σύστημα, ενισχύοντας την οργάνωση των παραγωγών τους. Είναι σημαντικό επίσης να διατηρήσουμε και να αναπτύξουμε περαιτέρω την κοινή οργάνωση αγοράς. Πιστεύουμε ότι χάρη στον κανονισμό δημιουργήθηκε μία άμεση σχέση παραγωγών και αγοράς χάρη στις οργανώσεις των παραγωγών και στις ενώσεις οργανώσεων παραγωγών. Χρειάζεται λοιπόν να αναπτυχθούν περαιτέρω αυτές οι δραστηριότητες και θα πρέπει να δώσουμε ίδια έμφαση στην διατήρηση της γεωργίας αλλά και στην πρόθεση της καινοτομίας. Επίσης, ε, να αναπτύξουμε πολιτικές πρόθεσης της ποιότητας, ε, προαγωγής ε, της παραγωγής, ανάπτυξη της καινοτομίας, πρόθεση της φιλοπεριβαλλοντικής παραγωγής, βιολογικής παραγωγής και ενίσχυση της συγκέντρωσης της προσφοράς. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε όλο μια ραγδαία αύξηση της ε, ζήτησης για βιολογικά προϊόντα. Θα πρέπει λοιπόν η αγορά να προσαρμοστεί στις νέες αυτές ε, τάσεις. Στη συνέχεια θα δούμε ποιες είναι οι σχέσεις των παραγωγών με τις μεγάλες αλυσίδες διανομής. Άρα από αυτή την άποψη θα πρέπει να επενδύσουμε και στην διαφύλαξη της ανταγωνιστικότητας ε, του κλάδου των απορροκυπευτικών. Και άρα στην πρόθεση της ποιότητας ε, με ειδικευμένο προσωπικό, με έμφαση στην καινοτομία και στις διαδικασίες και στα προϊόντα και στη λήψη υπόψη της περιβαλλοντικής διάστασης, γιατί η περιβαλλοντική αξία της ε, γεωργικής παραγωγής είναι επίσης σημαντική. Τώρα για την ανταγωνιστικότητα. Ρίχνοντας μια ματιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με 28 χώρες και διαφορετικά χαρακτηριστικά, διαπιστώνουμε ότι θα πρέπει να προσαρμόσουμε την κοινή οργάνωση αγοράς στις ιδιαιτερότητες των διαφόρων χωρών. Στον κανονισμό δεν χρειάζεται να έχουμε θετικούς ή αρνητικούς καταλόγους. Προτιμώ ένα γενικό πλαίσιο με μεγαλεπίβολες δράσεις που θα προσαρμοστούν στις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας. Θα πρέπει να αξιοποιηθούν τα ατού της Ευρώπης και με βάση τις ιδιαιτερότητες να προσδιορίσουμε τις απαιτήσει από κάθε χώρα. Έτσι θα μπορέσουμε με ένα μικρό, έστω και μικρό επίπεδο οργάνωσης να την καταστήσουμε πιο αποτελεσματική και να εφαρμόσουμε καλύτερα και την κοινή οργάνωση αγοράς. Ανακύπτουν εδώ δύο ερωτήματα. Τι γίνεται με τις χώρες που έχουν χαμηλό βαθμό οργάνωσης παραγωγής, οργάνωση παραγωγών. Θα πρέπει ε, να εφαρμόσουμε ένα, μια κοινή οργάνωση αγοράς ε, που θα προωθεί την περαιτέρω οργάνωση σε συνεταιρισμούς ώστε να διευκολυθεί καλύτερα η θέση σε εμπορία. Ένα Μια σταδιακή διαδικασία που θα λαμβάνει υπόψη τους διάφορους στόχους, τους περιβαλλοντικούς, την ανάγκη συγκέντρωσης της προσφοράς, η σταδιακή χρηματοδότηση, όλα αυτά θα επιτρέψουν την περαιτέρω ανάπτυξη των οργανώσεων παραγωγών. Διότι βεβαίως το χαμηλό επίπεδο οργάνωσης είναι αρνητικό και κάτι άλλο αρνητικό είναι ο πολύ μεγάλος αριθμός ε, <clears throat> συνεταιριστικών οργανώσεων που δεν μπορούν να προσαρμοστούν στην αγορά. 60% δηλαδή να υπάρξει επιδότηση για όλες τις οργανώσεις παραγωγών, τους συνεταιρισμούς. διότι ε, έχουμε παραμελήσει τη βοήθεια προς αυτές τις οργανώσεις. Πρέπει λοιπόν να διορθωθεί αυτή η κατάσταση. Πρέπει να ενισχύσουμε οπωσδήποτε το ρόλο των συνεταιρισμών αυτών, παραγωγών και για την ίδια την παραγωγή, τον τρόπο διάθεσης του προϊόντος στην αγορά και τη σχέση μεταξύ παραγωγής και διανομής, συλλογικές ενέργειες ε, για διαφήμιση συλλογικές ενέργειες για να αντιμετωπιστούν οι κρίσει για την έρευνα και την καινοτομία. Όλα αυτά είναι θεμελιώδη εργαλεία για να υπάρξει βελτίωση της κατάστασης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για τον Νότο ιδίω. γιατί θέλουμε να ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη και τη συσπήρωση αυτών των οργανώσεων για τη διατήρηση της κρίσης τώρα, για τη διαχείριση. Υπάρχουν οι συγκυριακές κρίσεις που μπορούν να είναι τμήματα των ε, λειτουργικών προγραμμάτων σε σχέση με τα προϊόντα και ο παρόν κανονισμός ε, δεν είναι συχνά επαρκής για να επιλύσει τα προβλήματα ακριβώς σε επίπεδο διαχείρισης. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να δημιουργήσουμε ένα κανονισμό, έναν μηχανισμό που να επιτρέπει να προσαρμοζόμεθα εύκολα στις αλλαγές στην αγορά για να βοηθήσουμε τους παραγωγούς του νότου της Ευρώπης να αποφεύγουν ένα τμήμα της παραγωγής τους να πηγαίνει χαμένο. Αυτό έχει συμβεί ιδίω στο νότο της Ευρώπης. Διότι ιδίω τα ευαίσθητα προϊόντα ορισμένε φορέ δεν υπάρχει δυνατότητα να διατεθούν και χάνονται, σαπίζουν. Τα, οι ντομάτε για παράδειγμα. Γιατί ορισμένα προϊόντα ε, είναι δύσκολο να διατηρηθούν. Αυτό είναι ένα συμπληρωματικό κίνδυνο. Άρα οι παρεμβάσει πρέπει να είναι ταχύτατε για να υπάρξει σωστή διαχείριση. Για το σύνολο τη παραγωγή. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή θα πρέπει να είναι μια προσπάθεια κοινή διαχείριση τη ε, κρίση που να επιτρέπει στι οργανώσει των παραγωγών και γενικά στην αλυσίδα παραγωγή και διανομή να αντιμετωπίζουν τι κρίσει, Να δώσουμε δηλαδή τη δυνατότητα να αποσυρθούν προϊόντα από την αγορά αν δεν υπάρχει δυνατότητα διάθεση πολύ σύντομα. Για παράδειγμα, όταν υπήρξε το εμπάργκο για τη Ρωσία ή το μικρόβιο ή κόλλη, τότε πρέπει να δίνονται δυνατότητες να αντιμετωπιστούν αυτές οι κρίσεις. Πρέπει να υπάρχει δηλαδή σωστή, σωστό κανονιστικό πλαίσιο. Διότι αν δεν υπάρχει αυτό, οι παραγωγοί προτιμούν να ε, θέσουν τα προϊόντα στην αγορά, έστω και με κίνδυνο να μην μπορέσουν να διατεθούν, παρά να κινδυνεύσουν να τα χάσουν τόσοι άλλους εάν ε, αποσυρθούν. Πρέπει λοιπόν να βρεθεί ένας μηχανισμός που να μας επιτρέπει να εγγυόμεθα στους παραγωγούς ένα συγκεκριμένο εισόδημα. Θα μπορούσε αυτό να γίνει και μέσω ενός συστήματος ασφαλίσεων ε, της παραγωγής. Δηλαδή ενδεχομένως να ασφαλίζεται συνολικά το σύστημα εμπορικής διάθεσης. Συχνά μας λένε ότι πρέπει να φτάσουν τα προϊόντα, τα προϊόντα μας και στις πιο απομακρυσμένες αγορές. Αλλά για να φτάσουμε σε αυτές τις ε, απομακρυσμένες αγορές ε, όπως η Κίνα, οι Ηνωμένε Πολιτείε, ιδίως για τις μικρότερες χώρες, αν δεν υπάρχει ένα καθεστώς ασφαλίσεων ή ε, αν ε, οι ασφαλείς πρέπει να καλύπτουν πολύ μακροχρόνια ταξίδια, τότε θα είναι πολύ ψηλά τα ασφάλιστρα ή δεν ασφαλίζουν καν ορισμένε εταιρείε. Πρέπει λοιπόν να βρεθεί τρόπος να ασφαλίζονται τέτοιε αποστολέ γιατί υπάρχουν και φυτο-υγειονομικές κρίσεις και εμπορικές κρίσεις, το είπαμε. Υπάρχουν στρεβλώσεις τη αγορά, ε, διακυμάνσει στην αγορά, διακυμάνσει των τιμών. Υπερβολικές πτώσεις των τιμών, για παράδειγμα. Εδώ πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα. Για παράδειγμα και πάλι το ρωσικό εμπάργο. Όταν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να υπάρχουν μέσα στο λειτουργικό πρόγραμμα συγκεκριμένες προβλέψεις και να ε, στοχεύονται επαρκώς οι επαρκείς πιστώσεις για να αντιμετωπιστούν αυτές οι κρίσεις. Γιατί έχει μεγάλη σημασία η ταχύτητα της παρέμβασης. Αν υπάρξουν διοικητικές καθυστερήσεις λόγω υπερβολικής γραφειοκρατίας δεν κάνουμε τίποτα. Αλλιώς ε, τα ίδια τα κράτη-μέλη δεν θα μπορέσουν να διαχειριστούν συνολικά τέτοιες κρίσεις. Τέλος, <clears throat> δωρεάν διανομή γεωργικών προϊόντων. Και αυτό είναι σημαντικό που έχει δώσει θετικά αποτελέσματα. Αλλά υπό την προϋπόθεση ότι θα πρέπει να γίνεται με συνεχή και προγραμματισμένο τρόπο. Ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν ευαίσθητα προϊόντα και αν δεν μπορεί να υπάρξει βιομηχανική μεταποίηση πρέπει να δίνουμε τη δυνατότητα στους συνεταιρισμούς ιδιαίτερα για προϊόντα λοιπόν πρέπει να καταναλωθούν σύντομα, να τα διαθέσουν, εάν δεν υπάρχει καμία άλλη δυνατότητα, να τα διαθέσουν δωρεάν. Και η εμπειρία που είχαμε φέτος, είχαμε αύξηση κατά 5% των προϊόντων που διατέθηκαν ε, δωρεάν, είναι θετική. Αυτό πρέπει να γίνει μόνιμο. Ε, τώρα έχουμε βεβαίως και τα περιβαλλοντικά μέτρα, αλλά δεν θα αναφερθώ, ε, θα μιλήσει ο Ζάκη αυτά. Θέλω τώρα να μιλήσω ε, για το νέο κανονισμό που είναι πολύ ικανοποιητικό για την διαφήμιση των προϊόντων. Είναι πολύ βασικό να έχουμε επαρκές πλαίσιο για την διαφήμιση και την προώθηση λοιπόν των προϊόντων μας ιδίως ε, για τα προϊόντα υψηλής ποιότητας, ε, τις ονομασίες ή ενδείξεις γεωγραφικής προέλευσης έχουν μεγάλη σημασία. Και πρέπει να γνωρίζει ο καταναλωτής ε, τα προϊόντα αυτά υψηλής ποιότητας για να μπορεί να τα αγοράσει. Για να ενδιαφερθεί για να τα αγοράσει. Δυστυχώς ακόμη δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση του κοινού για τέτοιου τύπου υψηλής ποιότητας προϊόντα ιδίως ε, στις νέες χώρες μέλη, όπου προσπαθούμε και εκεί να διαθέσουμε, να διατεθούν οι παραγωγές των νέων χωρών προς ε, μακρινές χώρες, για παράδειγμα Κίνα, Βιετνάμ. Πρέπει ε, να υπάρχει μια πλαισίωση αυτών των προσπαθειών εμπορίας των προϊόντων μας. Πολλές φορές το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι γνωστά αυτά τα προϊόντα ευραίως. Υπάρχει λοιπόν το πρόγραμμα που λέγεται ε, εκπαίδευση για την διατροφή στα σχολεία. Θα ήταν καλό να έχουμε και άλλα παρόμοια τέτοια προγράμματα, δεν είναι αρκετά εκτεταμένα. Ε, και Είναι λοιπόν βασικό να υπάρχει ε, εκπαίδευση ε, στα σχολεία για ε, να ενημερωθούν οι μαθητές και επίσης να ενημερωθούν για τα φρούτα και άλλα προϊόντα που είναι καλό να καταναλώνουν. Και ιδιαίτερα για να αντιμετωπίσουμε τις κρίσεις διάθεσης. Ένας άλλος τομέας που μας ενδιαφέρει είναι τα φυτο και οι συμφωνίες που υπάρχουν με τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Πιστεύουμε λοιπόν ότι η Ευρώπη πρέπει να βοηθήσει περισσότερο και την σύναψη διμερών συμφωνιών για να είναι πιο αμοιβαίε και για να έχουν όλοι τη δυνατότητα να εφαρμόσουν με το σωστό τρόπο τις διμερείς συμφωνίες. Αλλά παράλληλα πρέπει να υπάρχει και κάποια ομοιογένεια αυτών των συμφωνιών. Οι χώρες που θέλουν να εισαγάγουν ε, τέτοια προϊόντα στην Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίζονται ομοιογενώς και να βοηθήσουμε και τις ε, δικές μας χώρες ε, που θέλουν να εξαγάγουν. Με ομοιόμορφο τρόπο να εξάγουν για να αποτύχουμε τις εμπορικές αποτυχίες πολλές φορές σε αυτό το τομέα. Οπότε θα περάσω τώρα στην τελευταία διαφάνεια και μετά ο Ζακ θα αναφερθεί σε άλλες πλευρές του θέματος. Τι θέλω να πω. Από ό,τι βλέπετε, ο κανονισμός έχει περίπου ολόκληρο τον ίδιο στόχο. Έχει στόχο τη διατροφή, την προστασία του περιβάλλοντος και την ε, διατήρηση της υπαίθρου. Προσπαθούμε να προωθήσουμε την συμπληρωματικότητα μεταξύ αυτών των τριών στόχων. Για να γίνει αυτό πρέπει να έχουμε οικονομίες κλίμακας, να κάνουμε την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων, να δαπανίσουμε λιγότερα και να έχουμε λειτουργικά προγράμματα για τις ε, επαγγελματικές οργανώσεις πολύ πιο αποτελεσματικά. Τα λειτουργικά προγράμματα είναι ο καλύτερος τρόπος για την ανάπτυξη της αγοράς. Ευχαριστώ πολύ. Θα παραγώ τη σκητάλη για λίγα λεπτά για να επισημάνω δύο θέματα που κατά τη γνώμη μας είναι σημαντικά και για τον τομέα των απορροκυπευτικών και για τη στρατηγική μας αλλά και για την κοινή οργάνωση αγοράς απορροκυπευτικών ε, και τα επιχειρησιακά προγράμματα. Θα πω δύο λόγια και για το, την περιβαλλοντική διάσταση. Ήδη από το 2007 η κοινή οργάνωση αγοράς απορροκυπευτικών ε, συμπεριέλαβε στα μέτρα της και κάποια περιβαλλοντικά μέτρα και μάλιστα ήταν πραγματικά προπομπός ο κλάδος των απορροκυπευτικών και πρωτοστάτησε σε τέτοια περιβαλλοντικά μέτρα. Και αυτό επηρέασε και την παραγωγή και την κατανάλωση. Δηλαδή το θέμα των κλιματικών συνθήκων επηρεάζουν τον τομέα και σε επίπεδο παραγωγής και σε επίπεδο κατανάλωσης. Και το γεγονός ότι έχουμε πραγματικά μια δυναμική διαταραχή του κλίματος και κλιματικών αλλαγών, ε, έχουμε πολύ πιο έντονες περιόδους ανοβρίας ε, και πολύ ζέστη στις χώρες του Νότου, αλλά και περιόδους έντονων ε, βροχοπτώσεων, ε, αντίξεων καιρικών φαινομένων, ε, ανεμοστροβίλων, καταιγίδων. Οπότε οι αλλαγές του κλίματος δημιουργούν και προκλήσεις στους παραγωγούς των απορροκυπευτικών, αλλά ταυτόχρονα επηρεάζουν αρνητικά την παραγωγικότητα και την ποιότητα της παραγωγής. Γι' αυτό επήγει η πρόθεση της καινοτομίας και της εφαρμογής της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης προκειμένου να προσαρμοστούμε σε αυτές τις αλλαγές του κλίματος. Και επανέρχομαι σε αυτά που είπε ο συνάδελφος από το Πανεπιστήμιο Βάχενιγκεν. 10% είναι μόνο τα περιβαλλοντικά μέτρα σε σχέση με το σύνολο των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Θέλουμε όμως πιο ανοιχτά, πιο εγκάρσια, πιο σαφή και πιο ασφαλή περιβαλλοντικά μέτρα. Θα αναφερθώ σε μία πτυχή αυτού του θέματος. Στα πλαίσια των επιχειρησιακών προγραμμάτων, μόνο τα συμπληρωματικά μέτρα λαμβάνονται υπόψη. Θα ήταν καλύτερο και σαφέστερο ε, να ε, είναι επιλέξιμα τα επιρρεβλητικά μέτρα και να χρηματοδοτούνται στο σύνολό τους από τα επιχειρησιακά προγράμματα. Και ένα θέμα που θα πρέπει να επεξεργαστούμε περισσότερο στο μέλλον είναι κάποιες απώλειες ε, του εισοδήματος, γιατί έχουμε 25 ε, με 30% της παραγωγής που χάνεται από την ε, φάση της παραγωγής μέχρι την κατανάλωση. Επίσης, καινοτομία. Νευραλγικό σημείο και για το παρόν αλλά και για το μέλλον του κλάδου. Γιατί θα πρέπει συνεχώς να προσαρμόζουμε την παραγωγή στη ζήτηση και να βελτιώνουμε την ανταγωνιστικότητα του κλάδου. Και είναι γνωστό τη σπάση ότι υπάρχουν φαινόμενα στρέβλωσης ανταγωνισμού του κλάδου, κυρίως από τις τρίτες χώρες, αθέμητο ανταγωνισμό και προβλήματα λόγω των μη δασμολογικών φραγμών. Θα πρέπει λοιπόν να διατηρήσουμε και να μειώσουμε το κόστος παραγωγής, ταυτόχρονα διαφυλάσσοντας και βελτιώνοντας την ποιότητα. Και ίσως ε, ε, διευρύνοντας την παραγωγή, διαφοροποιώντας την για να τα αποκρίνεται στις ανάγκες και στη ζήτηση των καταναλωτών. Καινοτομία λοιπόν για τις νέες ε, αναζήτηση νέων ποικιλιών, για νέες τεχνικές πιο βιώσιμης προστασίας, νέες συσκευασίες, νέα προϊόντα που θα προσαρμόζονται καλύτερα στη, στο νέο τρόπο ζωής και στις νέες συμπεριφορές των καταναλωτών και μαζί με τη Φρέσφελ, που είναι μια οργάνωση αδελφή της Κόπα Κοζέκα δημιουργήσαμε λοιπόν μια ομάδα εργασίας για να προτείνουμε στα πλαίσια του ορίζοντας 2020 προτεραιότητες για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη για την επόμενη πενταετία και κυρίως για τα απορροκυπευτικά. Και φτάνουμε στα συμπεράσματα τώρα. Τι θα θέλαμε κατά κλείδι να τονίσουμε. Ε, βέβαια η έκθεσή μας θα αναφέρει πιο διεξοδικά. Καταρχήν να τονώσουμε την κατανάλωση πρώτα απ' όλα, γιατί μέσα σε 8-10 χρόνια, με βάση τις μελέτες του Φρέσφελτ, έχουμε χάσει περίπου 18% ε, καταστήματα, ε, μάλλον ε, ποσοστιαίες μονάδες κατανάλωσης στην Ευρώπη. Και έχουμε διάφορα προγράμματα για τα φρούτα στα σχολεία, για συνεργασία με τρίτες χώρες, ευαισθητοποίηση και ενημέρωση κυρίως των νέων για την ανάγκη της συμπερίληψης των απορροκευτικών στην διατροφή. Όλα αυτά τα μέτρα είναι πολύ σημαντικά για το μέλλον του κλάδου. Επίσης θα πρέπει να στηρίξουμε τις εξαγωγές μας προς τις τρίτες χώρες. Και να προσπαθήσουμε να γενικεύσουμε την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαιότητας, να ελαφρύνουμε ή να καταργήσουμε τους φυτογενομικούς φραγμούς και τους δασμολογικούς φραγμούς και τέλος να διατηρήσουμε, αυτό είναι ε, θεμελιώδους σημασίας, την κοινή οργάνωση αγοράς οπωροκυπευτικών. Γιατί όπως είπε ο κύριος Τρεντίνη, η κοινή οργάνωση αγοράς είναι πραγματικά προσανατολισμένη προς την αγορά, ενώ η παραγωγή και οι οργανώσεις των παραγωγών ε, εξαρτώνται από το εισόδημα που τους δίνει η αγορά και πολύ συχνά ε, ταλανίζονται είτε από διαρθρωτικές είτε από συγκυριακές κρίσεις που πλήττουν τον κλάδο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Ήταν ε, πολύ περιεκτικές οι ομιλίες σας. Τελικά είχαμε την πολυτέλεια του χρόνου και δεν χρειάστηκε να σας πιέσουμε να συντμήσετε τις παρουσιάσεις σας. Αλλά μας δώσατε πραγματικά πολύ σημαντικές πληροφορίες ε, για να αντιληφθούμε τις ιδιαιτερότητες ε, και τις ειδικές περιστάσεις του κλάδου των οποροκυπευτικών. Πρώτα θα δώσω το λόγο στον κύριο Μέλο που είναι ο εισηγητής μας. Ευχαριστώ Πρόεδρε να ευχαριστήσω τον κύριο Πόσμαν, Μπέιμαν για την παρουσίαση της κατάστασης στα βόρες στις βόρειες αλλά και τους ε, δύο επόμενους ομιλητές για τις νότιες χώρες. Αυτές οι εκθέσεις, ε, οι μελέτες είναι για μας πάρα πολύ σημαντικές. Η δική μου έκθεση είναι πολύ συγκεκριμένη αφορά τις οργανώσεις παραγωγών στον τομέα αυτό. Οπότε αυτές οι μελέτες πραγματικά είναι πάρα πολύ ωφέλιμες και χρήσιμες. Σημείωσα πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα λάβω υπόψη. Έχω κάποιες αμφιβολίες και κάποιες διευκρινήσεις που θα ήθελα να ζητήσω. Πρώτον, στον κύριο Μπέιμαν, σε ό,τι αφορά τους κανόνες στις ε, συστάσεις, αναφέρεται ότι η παραγωγοί της Βόρειας Ευρώπης δεν ζητούν καινούριους κανόνες, ζητούν απλοποίηση των υφιστάμενων κανόνων. Σας ερωτώ πώς είναι δυνατόν να επιτύχουμε το ένα χωρίς το άλλο, δηλαδή πώς είναι δυνατόν να ε, απλοποιήσουμε το νομοθετικό πλαίσιο χωρίς να το αλλάξουμε. Ποια είναι η, η έννοια αυτής της απλοποίησης λοιπόν. Δεύτερον, Σε ό,τι φορά την ε, περιγραφή των οργανώσεων παραγωγών στο βορρά και το νότο. Ε, από ό,τι φαίνεται έχουμε μια τάση λιγότερων οργανώσεων παραγωγών αλλά ε, μεγαλύτερου μεγέθους. Υπάρχει κάτι το οποίο δεν κατάλαβα πολύ καλά διότι έτσι κι δεν έχω διαβάσει τη λεπτομέρεια των εκθέσεων αλλά Ε, έχουμε κάποια στοιχεία για τη γύραση του συστήματος στην ε, Ευρώπη. Ε, ε, στατιστικά έχουμε το εξής. Στην Ευρώπη έχουμε αυτή τη στιγμή ε, ένας γεωργός κάτω των 35 ετών για κάθε 9 γεωργούς άνω των 55. Ένας κάτω των 35 για κάθε 9 πάνω από 55 ετών. Σε ορισμένε χώρε του Νότου τη Ευρώπη, αλλά και στο Ηνωμένο Βασίλειο, που δεν είναι Νότια Ευρώπη, ε, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, αλλά και Ηνωμένο Βασίλειο και η Βουλγαρία, σε αυτέ τι χώρε έχουμε ένα γεωργό με ηλικία κάτω των 35 ετών για κάθε 20 ηλικία άνω των 55. Ακόμα χειρότερη δηλαδή η αναλογία. Στην Πολωνία, την Αυστρία και την Γερμανία η κατάσταση είναι λίγο διαφορετική. Ένας γεωργός κάτω των 35 για κάθε τρεις άνω των 55. Πολωνία, Αυστρία, Γερμανία λοιπόν βρίσκονται σε λίγο καλύτερη στατιστικά κατάσταση, αλλά και πάλι η κατάσταση είναι ανησυχητική. Υπάρχει μια γύρανση του ε, παραγωγικού εστού στην Ευρώπη. Αυτό αντικατοπτρίζεται ε, και στο κλάδο των φρούτων και προεκπαιδευτικών. Και μήπως θα έπρεπε να έχουμε μια εκπαιδευτική πολιτική προσαρμοσμένη σε αυτό το πρόβλημα. Μετά, μια επόμενη ερώτηση για τον κύριο Τρεντίνη και τον κύριο Ντάσκ για τις χώρες της Νότιας Ευρώπης που έχει σχέση με μια πρόσφατη πολιτική απόφαση να ανοίξει ε, η αγορά της Ευρώπης ε, σε ορισμένες χώρες της Βόρειας Αφρικής. Ε, στη Βόρεια Αφρική η παραγωγή είναι η ίδια και την ίδια μάλιστα εποχή με τις χώρες της Νότιας Ευρώπης, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία κυρίως. Έχει ε, εντοπιστεί, έχει παρατηρηθεί κάποια συνέπεια η ε, αυτής της απόφασης στην αγορά. Τώρα, κάτι άλλο. Σχέση ανάμεσα στους οργανώσεις παραγωγών με τις ε, διόδους, με τα κανάλια εμπορίας. Ε, μερικές φορές, πολλές φορές, είναι πολύ δύσκολο ο παραγωγός να πουλάει το προϊόν, του με δίκαιο τρόπο, γιατί ε, ε τιμές υφίστανται πίεση προς τα κάτω, συμπιέζονται εξαιτίας των καλαλιών εμπορίας. Οπότε, πολιτικά θα μπορούσαμε ή θα έπρεπε να λάβουμε μέτρα προκειμένου να ρυθμίσουμε τη σχέση ανάμεσα στους παραγωγείς, στην παραγωγή και τη διανομή. Έτσι ώστε οι παραγωγοί να απολούν το προϊόν τους με έναν τρόπο δίκαιο. Επίσης θα ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε παρατηρήσει σε σχέση με τους συνεταιρισμούς μια δυσκολία η οποία προκύπτει από κάποιο ρασιτεχνισμό στη διαχείριση των συνεταιρισμών. Πολλές φορές δηλαδή οι γεωργοί δημιουργούν οργανώσεις παραγωγών και οι οργανώσεις αυτές πρέπει να λειτουργούν ε, ως πραγματικές επιχείρησεις. ανταγωνίζονται μεταξύ τους άλλωστε. Το είπε ο Μπέιμαν για παράδειγμα. Είναι μερικέ ε, εκμεταλλεύσει που γίνονται τόσο μεγάλε που προτιμούν να μην μπουν σε οργανώσει παραγωγών και να λειτουργήσουν αυτόνομα. Ανταγωνιστικά με του οργανώσει παραγωγών. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται επαγγελματισμό. Υπάρχουν πολλέ οργανώσει, ή κάποιε τουλάχιστον, που δεν είναι κερδοφόρε, όχι γιατί δεν έχουν καλή θέληση, όχι δεν δουλεύουν, αλλά γιατί δεν δουλεύουν επαγγελματικά. θα έπρεπε να δώσουμε κάποια κίνητρα για την επιμόρφωση των στελεχών τους ε, και για την ε, πρόσληψη επαγγελματιών managers για να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Θα, με, θα ήταν πολύ ωφελή μια, μια απάντηση από εσά για μένα. Επίσης, καταγράφω τη σημασία που δίνεται στην πολιτική διανομής φρούτων και προκυπευτικών στα σχολεία. Πολύ συχνά μιλάμε για τα πλεονεκτήματα της μεσογειακής ε, διατροφής. Εμείς δεν είμαστε Μεσόγειο στην Πορτογαλία, αλλά το συμμεριζόμαστε. Οπότε, ε, έχει νόημα να ακολουθήσουμε πολιτικές αλλαγές των διατροφικών ε, συνηθιών από παιδαγωγικής πλευράς χρειάζεται να ακολουθεί μια τέτοιου είδους πολιτική αλλαγής διατροφικών συνθήκων παράλληλα με τη διανομή φρούτων και απορροκυπευτικών. Επίσης, σε ό,τι αφορά τον νότο της Ευρώπης, την αντιμετώπιση των κρίσεων ε, και το πώς οι οργανώσεις παραγωγών μπορούν να βοηθήσουν. Έχετε κάτι πιο συγκεκριμένο να μου πείτε. Ευχαριστώ. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες αυτές τις παρουσιάσεις. Σας ευχαριστούμε. Ήδη καταλαβαίνω ότι αρχίσατε κιόλα να εμπλουτίζετε και να αναπτύσσετε την έκθεση. Ε, Ο κύριος Γλέζος. Κύριε Γλέζο, έχετε το λόγο. Αρκετά ενδιαφέρουσες οι εισηγήσεις και πολύ σημαντικές. Όμως δημιουργούν δύο προβλήματα δημιουργούνται. Καταρχήν ο παραγωγός θεωρεί στο συνεταιρισμό που βρίσκεται ότι υπάρχουν μεγάλοι ανταγωνιστές του οι οποίοι τον συντρίβουν. Τους λέει εχθρούς, τους λέει αντιπάλους, ανταγωνιστές. Όπως και να τους πούμε είναι τα μεγάλα καρτέλ τα οποία του αρπάζουν την παραγωγή και συντρίβουν το μικρό παραγωγό. Ερώτημα. Ποια είναι η πολιτική της Κομισιόν, ποια είναι η πολιτική της ε, Ευρωπαϊκής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μας για να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Το δεύτερο, ανάμεσα στον παραγωγό και στον καταναλωτή υπάρχει ο μεσάζων, υπάρχει ο έμπορος. Αυτός είναι ο κερδισμένος, αυτός είναι που κερδίζει τα πάντα. Τελευταία έχει αποκαλυφθεί ότι η απόσταση ανάμεσα στο προϊόν που, καταναλών, που παράγεται και καταναλώνεται ο έμπορας κερδίζει τα περισσότερα το κερδίζει αφάνταστα ποσά πως αντιμετωπίζεται το πρόβλημα αυτό το τεράστιο και επειδή είμαστε τώρα όπως έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες σε αλκιονίδες μέρες και βλέπουμε να ανθίζουν να ξεγελιώνται οι αμυγδαλιές και να ανθίζουν θα έλεγα μέσα από αυτό το πλαίσιο των εισηγήσεων που δημιουργούν μια ατμόσφαιρα αλκιονίδων ημερών να μην παρασυρθούμε κι εμείς από τις διάφορες τοποθετήσεις και ξεχάσουμε την πραγματικότητα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Γλέζο. Ο κύριος Ροπέ. Ε, Ευχαριστώ πολύ για τις παρουσιάσεις που κάνατε. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσες και χρήσιμες. Είστε όντως ε, ειδικοί ο καθένας στον τομέα του. Είμαι Λιθουανός όπου είναι πολύ χαμηλή η οργάνωση, το ποσοστό οργάνωσης των παραγωγών. Ξέρετε, στη Σοβιετική εποχή ήμασταν υποχρεωμένοι να συμμετέχουμε σε συνεταιρισμούς και γι' αυτό τώρα πολλοί έχουν ένα ψυχολογικό φραγμό λόγω αυτής της, ε, του καταναγκασμού. Θεωρούν ότι η συνεργασία μεταξύ παραγωγών είναι κάτι αρνητικό. Θέλω λοιπόν να θέσω το εξής ερώτημα. Αν θυμάμαι καλά αναφέρατε ότι η παραγωγή φρούτων και λαχανικών έχει μειωθεί, συγγνώμη, η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών έχει μειωθεί κατά 18% στην Ευρώπη. Ε, μπορείτε να μου δώσετε λόγους γι' αυτό. Ο πρώτος ομιλητής αναφέρθηκε λοιπόν στους συνεταιρισμούς, ε, τη συνεργασία των παραγωγών. Σε ποιο επίπεδο πρέπει να γίνεται συνεργασία. Ποιο είναι το πιο κατάλληλο επίπεδο. Θα πρέπει να συμμετέχουν μόνο οι πρωτογενείς παραγωγοί, αυτοί ακριβώς που παράγουν τα προϊόντα, ή θα πρέπει να υπάρχει μια οργάνωση που να ε, συμπεριλαμβάνει και τους διανεμπόρους ούτως ώστε να υπάρχει δίκαιη κατανομή του κέρδους. Είπατε επίσης ότι οι οργανώσεις παραγωγών και οι συνεταιρισμοί γίνονται όλο και μεγαλύτεροι. Έχετε στατιστικά στοιχεία. Σε ποιους τομείς διαπιστώνουμε τα μεγαλύτερα ποσοστά συγκέντρωσης. Στις χώρες όπου το ποσοστό οργάνωσης ε, συμμετοχής στους συνεταιρισμούς είναι μεγαλύτερο ή στις χώρες όπου είναι μικρότερο. Επίσης, ανεξάρτητα από το είδος των παραγωγών, το βασικό είναι να είναι δίκαια οργανωμένοι και διαρθρωμένη αλυσίδα παραγωγής και διανομής. Θεωρείτε ότι χρειάζεται δεσμευτικός κανονισμός για τη σχέση μεταξύ παραγωγών, ε, μεταποιητών και ε, για λιανεμπορίου. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Δεκάστρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ Πολύ σύντομα γιατί θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους ε, εμπειρογνώμονες και προσκεκλημένους μας. Μας έδωσαν ένα πολύ καλό και συγκεκριμένο πλαίσιο για να καταλάβουμε τις δυσχέρειες αλλά και τις ευκαιρίες, τις σημαντικές ευκαιρίες ε, που υπάρχουν για βελτίωση της κατάστασης σε αυτό το τομέα. Ακούσαμε πρόσφατα για τις δυσχέρειές τους, ε, ακούσαμε για το ρωσικό εμπάργο και βεβαίως επηρεάστηκε πολύ ο τομέας των οποροκυπευτικών από αυτό το εμπάρκο και επίσης ε, η κατανομή των πόρων ε, της Κομισιόν στις διάφορες χώρες δεν είναι ιδανική. Να είμαι όμως σύντομος. Με βάση τα σχόλια που έχουν γίνει και τα αποτελέσματα που έχουμε επιτύχει, σίγουρα μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έχει υπάρξει κάποια βελτίωση τόσο στο βορρά όσο στο νότο. Ε, έχει υπάρξει βελτίωση του επίπεδου οργάνωσης, ε, όχι ίσως όσο ταχεία θα θέλαμε, αλλά παρόλα αυτά. Ερώτηση λοιπόν. Θεωρείτε ότι πρέπει να αναθεωρηθούν οι κοινέ οργανώσει αγορών οποροκυπευτικών και αν ναι, προ ποια κατεύθυνση. Γιατί από ό,τι βλέπω, καλά πάντα πράγματα, θα μπορούσαμε να τα βελτιώσουμε περαιτέρω αλλά εγώ δεν βλέπω ανάγκη για ριζική ε, μεταρρύθμιση των απορριπευτικών, των κοινών οργανώσεων αγορών του δηλαδή. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ. Και εγώ επιβεβαιώνω αυτά που μόλις είπε ο κύριος Δεκάστρο. Και εγώ δεν βλέπω να υπάρχει ανάγκη ριζικής μεταρρύθμισης των κοινών οργανώσεων αγορών του τομέα αυτού. Συγκεκριμένη ερώτηση όμως για τον κύριο Τρεντίνη η διαχείριση κρίσεων. Ήσασταν ιδιαίτερα επιφυλακτικός όσον αφορά τις δυνατότητες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σοβαρές κρίσεις, όπως η πολιτική κρίση που αντιμετωπίζουμε τώρα. Εγώ είμαι κάπως πιο αισιόδοξο. Εγώ νομίζω ότι οι οργανώσεις παραγωγών έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν ακόμη και μεγάλης κλίμακας κρίσης, όχι βέβαια τις χειρότερες, Όταν βλέπουμε πόσο αποδίδουν οι χρηματοδοτήσεις μας, πρέπει να κάνουμε διακρίσεις μεταξύ των οργανώσεων παραγών που έχουν ακριβώς δυνατότητα να αντιμετωπίσουν κρίσεις, έχουν τους αναγκαίους χώρους αποθήκευσης των προϊόντων, που έχουν δυνατότητα να μεταποιήσουν προϊόντα, αναφερόμεθα κυρίως στα φρούτα τώρα, και, γιατί ο μόνος τρόπος να ε, βγάλουμε από την αγορά ένα σημαντικό ε, ποσοστό της παραγωγής φρούτων είναι να τα μεταπίσουμε. Δεν νομίζω ότι η διανομή δωρεάν στους καταναλωτές είναι λύση. Διότι με χαρά ε, αγοράζουν, με χαρά δέχονται δωρεάν φρούτα και λαχανικά, αλλά αυτό δεν αυξάνει το εισόδημα των παραγωγών. Δεν θα συνηθίσουμε μετά να τα αγοράζουν. Επίσης, ε, σημαντικό ρόλο θεωρώ ότι θα παίξει το περιβάλλον και η προστασία του. Γιατί, για παράδειγμα, η χρήση εντομοκτώνων ε, πρέπει οπωσδήποτε να επανεξεταστεί στον τομέα αυτό των οποροκυπευτικών. Η έρευνα που γίνεται για τα θέματα αυτά μας δίνει πολύ διαφορετικές δυνατότητες ε, με βάση τις βέλτιστες πρακτικές για τον κλάδο αυτό. Πιστεύω λοιπόν ότι μέσω των λειτουργικών προγραμμάτων μπορούμε να αναπτύξουμε περαιτέρω τον τομέα αυτό που είναι σημαντικός για τους Γιώργους μας. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ντελαέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και τους καλεσμένους μας, τους ειδικού για τις παρουσιάσεις που μας έκαναν. Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε το λόγο για τον οποίο προωθούμε τις οργανώσεις παραγωγών. Ε, κυρίως για να διαφυλάξουμε το γεωργικό εισόδημα, το εισόδημα του παραγωγού. Τι γνώμη έχετε για τις σχέσεις μεταξύ παραγωγών, οι οργανώσεων παραγωγών και των ε, αλυσίδων διανομής. Ή μήπως θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τους κανόνες ανταγωνισμού για να επιτρέψουμε μια επανισορρόπηση της αγοράς και του σχετισμού δυνάμεων μεταξύ των μεγάλων αλυσίδων διανομής, των σούπερ μάρκετ και των παραγωγών μέσω των οργανώσεών τους. Και υπό το φως της κρίσης που βιώσαμε τα τελευταία χρόνια για το σχερίδια κόλλη το 2011 και πρόσφατα την κρίση που δημιουργήθηκε από το ρωσικό εμπάργκο, πώς ε, είναι δυνατόν να, ε, να φανταστούμε ότι ένα τμήμα της παραγωγής, όσο οργανωμένη και είναι, και είδαμε από τις ομιλίες σας ότι το επίπεδο οργάνωσης διαφέρει από χώρα σε χώρα. Πώς μπορούμε χάρη σε αυτό να ανατάξουμε τις αγορές χωρίς να έχουμε μαζική συσπήρωση των παραγωγών. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να μεταρρυθμίσουμε ή όχι την κοινή οργάνωση αγοράς, αλλά σίγουρα μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση με καλύτερη οργάνωση των παραγωγών. Των ανοργάνωτων εντός εισαγωγικών παραγωγών. Βέβαια, δεν νομίζω ότι ευσταθεί το να λέμε ότι όσοι δεν είναι σε συνεταιρισμούς ή οργανώσεις είναι ανοργάνωτοι, γιατί υπάρχουν μεγάλες δομές παραγωγής που έχουν τα δικά τους ε, ε, κυκλώματα διανομής ε, και διαχείρισης τη παραγωγής. Πάντως με τις κρίσεις που βιώσαμε τα τελευταία χρόνια στα προεκλογικά, θα, χρειαστεί να συσπηρώσουμε όλες τις εμπορικές δυνάμεις σε πρώιμο επίπεδο ώστε να περιορίσουμε τις απώλειες και τις ζημίες για τους παραγωγούς και να διορθώσουμε και την φθήνουσα πορεία που έχει πάρει η κατανάλωση απορροκυπευτικών. Γιατί υποχρηματοδοτείται η εκστρατεία πρόθεση. και στον κανονισμό για την πρόθεση θα πρέπει ίσως να βάλουμε κάποια νέα θεμέλια για να προωθήσουμε περισσότερο την κατανάλωση απορροκυπευτικών. Αυτές ήταν οι δικές μου σκέψεις για το θέμα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σεμπάστια. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τους ε, καλεσμένους μας. Πολύ ενδιαφέρουσες οι παρουσιάσεις ε, και πολλά διδαχθήκαμε από αυτές, αλλά μετά τη τελευταία παρέμβαση άρχισα να προβληματίζομαι και να ανησυχώ, γιατί μίλησε για το άνοιγμα των συνόρων και για τη μείωση των δοσμολογικών φραγμών και την κατάργησή τους για την καλύτερη πρόθεση των προϊόντων. Όπως είπε ο εισηγητής μας ο κύριος Μέλο, πολλά προϊόντα οπωροκυπευτικά παράγονται στη Βόρεια Αφρική την ίδια χρονική στιγμή με την παραγωγή στη Νότια Ευρώπη. Υπάρχουν όμως μεγάλες διαφορές στους όρους παραγωγής, περιβαλλοντικούς, υγειονομικούς, κοινωνικούς. Άλλες είναι οι συνθήκες παραγωγής στη Βόρεια Αφρική και άλλες στη Νότια Ευρώπη. Δεν υπάρχει ισότητα συνθήκων και όρων παραγωγής. Γιατί έχουμε υψηλέ κοινωνικέ, περιβαλλοντικέ, εργασιακέ απαιτήσει από του δικού μα ευρωπαϊκού παραγωγού για μια υφόρο γεωργία και είναι σωστό αυτό και εύστοχο, αλλά δεν πληρούνται οι ίδιε προποθέσει στην παραγωγή τη Βορειοαφρική. Οπότε δημιουργείται de facto ένα αθέμητο ανταγωνισμό με ολέθριε συνέπειε για του δικού μα παραγωγού. Και είναι σαφές αυτό που είπε ο κύριος Μέλλο, ότι έχουμε απερίμωση της υπαίθρου, εγκατάλειψη των γεωργικών δραστηριοτήτων ε, και εγώ στη Βαλένσια, στην Ανατολική Ισπανία, που είναι περιοχή που παραδοσιακά είχε μεγάλη γεωργική παράδοση, αυτή τη στιγμή απειλείται η ίδια η επιβίωση της γεωργίας. Εγκαταλείπονται χωράφια αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Εξαιτίας ε, του κατακλυσμού των αγορών μας ε, από φθηνά προϊόντα τρίτων χωρών που δεν πληρούν τις ίδιες υψηλές δικές μας ποροδιαγραφές. Οπότε μιλήσατε για άνοιγμα των συνόρων και κατάργηση των δασμών για να βελτιωθούν οι εισαγωγές, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι ε, κατάλληλο μέτρο. Θα το χαρακτήριζα ως και επικίνδυνο, αν κατάλαβα τουλάχιστον καλά την πρότασή σας. Σας ευχαριστώ, κυρία Πετήρ. Ε, ε, ε. Ευχαριστώ για αυτές τις τρεις παρουσιάσεις. Η μελέτη που μας παρουσιάσατε αφορά την περίοδο μέχρι το 2014. Στην, με τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ η κοινωνία αγοράς ξελίχθηκε ενισχύοντας την δυνατότητα δημιουργίας οργανώσεων παραγωγών ε, και ενώσεων οργανώσεων παραγωγών. Και επίσης ε, βελτιώθηκε η διαπραγματευτική ικανότητά τους. Ε, έχετε καταγράψει τις εξελίξεις αυτές που παρήχθησαν μετά την μεταρρύθμιση του 2014. Ευχαριστώ. Και τώρα ο λόγος στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Σάπς. Παρακαλώ. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που διοργανώσατε αυτή την πολύ, αυτό το πολύ ενδιαφέρον εργαστήριο για τον τομέα των προεκπαιδευτικών. Όπως γνωρίζετε και εμείς ε, εξετάζουμε αυτή την περίοδο τα αποτελέσματα της εφαρμογής της ε, μεταρρύθμισης του 2007. Και δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονό ότι καταλήγουμε σε παρόμοια συμπεράσματα με ορισμένα τουλάχιστον από ε, τα πορίσματα των μελετών. Είναι σαφές ότι ο κλάδος είναι ε, πολύ σημαντικός για την ευρωπαϊκή γεωργία. Είναι επίσης ένας πολύ δυναμικός κλάδος που έχει εξελιχθεί προς πολλές κατευθύνσεις προς την κατεύθυνση της συνεργασίας, της ε, ε, οργάνωσης της παραγωγής των παραγωγών, αλλά και προς την κατεύθυνση της εμπορίας των προϊόντων στα διάφορα κράτη-μέλη και πώς γίνεται αυτή. Για την ε, της Ευρωπαϊκής, Κομισιόν, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πολύ καλό που αυξήθηκε η συνεργασία και ο βαθμός οργάνωσης, όπως αναφέρθηκε και στις μελέτες. Η πρόοδος είναι αργή ενδεχομένως, ενδεχομένως υπερβολικά αργή σε ό,τι αφορά ορισμένους παράγοντες, αλλά υπάρχει, υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι ο βαθμός συνεργασίας και οργάνωσης αυξάνεται. Το άλλο σημαντικό στοιχείο είναι το εξής. Όπως γνωρίζετε, ε, το παρόν σύστημα προσφέρει δυνατότητες οι οποίες έχουν ε, τύχη εκμετάλλευση. Τα 24% των δαπανών μας ήταν σε περιβαλλοντικά μέτρα, για παράδειγμα. Αυτό είναι πολύ καλή πρόοδο. Ίσως μπορούμε να βελτιώσουμε την υλοποίηση, αλλά και αυτό νομίζω είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Μια πολύ σημαντική πτυχή απορρόφησης Οι βασικές αδυναμίες κατά την άποψή μας είναι η περιπλοκότητα του συστήματος και γενικότερα τα σχετικά με το ε, ε, νομικό περιβάλλον. ο τομέας των απορριπευτικών θα αποτελέσει τμήμα της ε, διαδικασίας απλοποίησης της κοινωνικής νομοθεσίας η οποία πιστεύουμε θα ολοκληρωθεί μέσω ε, εφαρμοστικών ε, και κατεξιοδότηση πράξεων κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους. Δεν μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα έτσι βέβαια, αλλά νομίζω ότι με την απλοποίηση θα μπορέσουμε να εδραιώσουμε το νομικό πλαίσιο ε, και να το κάνουμε πιο ευανάγνωστο, πιο εύκολα εφαρμόσιμο. Ακούσαμε τις ε, συστάσεις ε, των μελετών ε, και θα τις συμπληρώσουμε με τις απόψεις των κρατών μελών στο Συμβούλιο τα επόμενα δύο χρόνια. Με βάση όλες αυτές τις παρατηρήσεις ενδεχομένως θα τροποποιήσουμε το κανονιστικό πλαίσιο της αγοράς. Γνωρίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει κάποια στιγμή να υποβάλει κάποια πρόταση το 2018 το αργότερο. Αν θεωρήσουμε ότι είναι απαραίτητο, θα περιλάβουμε κάποια πράγματα και για τον τομέα των προκυπευτικών. Τώρα, έχουμε κάποιες ανησυχίες σε ό,τι αφορά την οικονομική διαχείριση. Γνωρίζετε ότι η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού ε, εξέτασε τη Δευτέρα το θέμα των προεκπαιδευτικών και υφίστανται ε, προγράμματα δράσης σε κάποια κράτη-μέλη στα οποία χρειάστηκε να παρέμβουμε προκειμένου να μειωθεί το ποσοστό σφαλμάτων και το πετύχαμε. Τα κράτη-μέλη προέβησαν σε διορθώσεις και απλοποίησεις. Επίσης, διαχείριση κρίσεων. Εξεπλάγημεν αυτό που, από αυτό που συνέβη με το ρωσικό εμπάργκο. Όμως νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Σύστημα του τελευταίους δύο μήνες ε, κατάφερε να αποσύρει πάνω από 600.000 τόνους από την αγορά. Με τα μέτρα, ε, έκτακτα μέτρα στήριξης. Ε, εξακολουθούμε να παρακολουθούμε την κατάσταση. Οι υπηρεσίε κομισιών έχουν σκοπό να συμμετάσχουν, να συνεχίσουν να συμμετέχουν ενεργά στη συζήτηση για τον κλάδο. Ε, ευχαριστούμε πολύ που μας δόθηκε ευκαιρία να σας ενημερώσουμε για τις απόψεις μας, ε, να ανταλλάξουμε γνώμες με όλους όσοι θέλουν να ε, σημειώσουμε πρόοδο. Περιμένουμε, να μένουμε με ενδιαφέρον τη συνεργασία του επόμενου μήνε. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Και τώρα οι εμπειρογνώμονές μας, αλλά παρακαλώ επιγραμματικά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριοι βουλευτές, για τις πολύ ενδιαφέρουσες και αναλυτικές ερωτήσεις. Δεν ξέρω αν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες όλων των ερωτήσεων, αλλά να απαντήσω στα κύρια θέματα που θέσατε. Λοιπόν, λοιπόν, που τα έχω. Ιδιαίτερα αυτά που είπε ο κύριος Μέλου ρώτησε πώς μπορούμε να απλοποιήσουμε τους κανόνες χωρίς να τους αλλάξουμε. Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Ε, άμα απλοποιήσεις κάπως θα αλλάξεις κιόλας. Τώρα δεν είναι δική μου δουλειά να προτείνω πολύ αναλυτικές ε, λύσεις. Αλλά από ό,τι κατάλαβα από τις εθνικές αρχές και εκπροσώπους του κλάδου ιδιαίτερα για τα περιβαλλοντικά μέτρα υπάρχει επαρκής πολυπλοκότητα. Εδώ τουλάχιστον θα μπορούσε κάτι να γίνει. Και αυτό το βλέπω και στις μελέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που περίχαν συνοψίσεις εθνικών αποτιμήσεων και δεν θεωρήθηκαν πολύ αποτελεσματικά όλα τα περιβαλλοντικά μέτρα. Και το καταλαβαίνω αυτό. Γιατί στον κλάδο αυτό υπάρχει, ε, υπάρχουν πολλές απαιτήσει για υψηλής ποιότητας ε, προϊόντα, υψηλής ποιότητας διαδικασία παραγωγής και αυτή προέρχεται από τα σούπερ μάρκετ, από τους καταναλωτές. Υπάρχει λοιπόν πολύ πίεση από αυτούς τους παράγοντες της αγοράς για να βελτιωθεί η περιβαλλοντική επίπτωση της παραγωγής των προϊόντων εδώ, λοιπόν μπορεί να υπάρξει κάποια απλούστευση. Επίσης, η εμπορία, η προώθηση των προϊόντων πρέπει να ενταθούν αυτός ήταν ο αρχικός μας στόχος. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη δυνατότητα των παραγωγών να διαθέτουν σωστά, να προωθούν τα προϊόντα τους στην αγορά. Και επίσης η καινοτομία και το ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό είναι επίσης πολύ ενδιαφέρον. Το θέσατε. Πώς θα βελτιώσουμε τον τρόπο λειτουργίας των συνεταιρισμών. Χρειάζεται εκπαίδευση, κατάρτιση, βοήθεια Νομίζω ότι όλοι οι συνεταιρισμοί και κατά συνέπεια όλοι οι παραγωγοί οπωσδήποτε θα ωφελούνταν από τέτοια πλαισίωση. Θα πρότεινα λοιπόν ε, να ασχοληθούμε περισσότερο με αυτούς τους τομείς. Φυσικά η παραγωγή είναι όλο και γυρεότερη και σε ορισμένες χώρες ε, η πλειονότητα είναι πάνω από 40 και πάνω από 50. Σαφή στάση. Ορισμένες εκμεταλλεύσεις ε, μόνο εν μέρη μπορούν να λειτουργήσουν και ορισμένες απλώς εγκαταλείπονται. Και οι νέοι που μένουν έχουν θέματα εκπαίδευσης. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Σε πολλές από τις ε, σχολές που προσφέρουν μαθήματα για διαχείριση επιχειρήσεων, για management. Δεν ε, αναφέρεται τίποτα για διαχείριση συνεταιρισμών γεωργών. Και στο δικό μου πανεπιστήμιο κανένα πρόγραμμα σπουδών δεν ασχολείται με την γεωργική παραγωγή. Κάπου επανέρχονται και χαίρομαι γι' αυτό στα εκπαιδευτικά προγράμματα, αλλά θα έπρεπε να υπάρχουν σε πολύ ευρύτερο βαθμό και δεν αλλάζουν εύκολα αυτά, ξέρετε. Πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο. Ναι, ναι, να τελειώνω μου είπατε. Μάλιστα, μάλιστα. Δηλαδή να καταλάβουν οι παραγωγοί ότι πολλά έχουν να από τους εταιρισμού. Πολλά άλλα θέματα αφορούν το ρόλο των παραγωγών στην αλυσίδα διάθεσης γεωρικών προϊόντων. Μα φυσικά είναι σημαντικός ο ρόλος τους. Πρέπει λοιπόν να ενισχυθεί και ο ρόλος σου σε όλη αυτή την αλυσίδα, στην αγορά. Και θα πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά τις διαστάσεις των ε, συνεταιρισμών. Θέλουμε να τις βοηθήσουμε ε, πέρα από οποιοδήποτε διάσταση να μεγαλώνουν. Ε, αυτά γιατί βλέπω ότι με κοιτάζει απειλητικά ο Πρόεδρος. Ο κύριος Τρεντίνη. Ευχαριστώ. Ήταν ε, πληθώρα των, ε, πληθώρα ερωτήσεων και πολύ ενδιαφέρουσες. Καταρχήν, ε, το θέμα των προϊόντων της Αφρικής. Για μένα είναι σημαντικό το θέμα της αμοιβαιότητα. Και όσο ετοίμαζα την παρουσίασή μου, εξέτασε την εξέλιξη του πληθυσμού μέχρι το 2050. Διαπιστώνουμε ότι σε όλες τις χώρες του κόσμου είχαμε ποσοστία μείωση. Παρόλο που μέχρι το 2050 ε, θα έχουμε αύξηση μικρή του πληθυσμού, η μόνη χώρα που θα διπλασιάσει τον πληθυσμό της είναι η Αφρική. Η μόνη Ήπειρος που θα διπλασιάσει τον πληθυσμό της από 890 εκατομμύρια θα περάσει στο 1,8 δισεκατομμύρια. Και μάλιστα πρόσφατα είχαμε ένα πρόγραμμα ε, και μία εμπορική αποστολή στην Τινησία. Αποφασίσαμε λοιπόν να μην θεωρήσουμε ως ε, στρατηγική ήπειρο την Ευρώπη, αλλά την Αφρική. Πρόσφατα, πριν από λίγα χρόνια, ασχοληθήκαμε με τις κινέζικες ντομάτες. Και Πολύ είπαν ότι θα εξαφάνιζε τις ντομάτες στην Ευρώπη. Όμως έχει αυξηθεί τόσο η κατανάλωση ντομάτας στην Κίνα, που η Κίνα πια δεν εξάγει τις ντομάτες της. Οπότε λύθηκε η απειλή από τις κινέζικες ντομάτες ε, που δεν κατακλείζουν πια την Ευρώπη. Υπήρξε μια αυτορύθμιση. Θα πρέπει να δούμε πού θα αυξηθεί ο πληθυσμός, γιατί εκεί είναι ελκυστικές αγορές που μπορούμε να διαχειοτεύσουμε τα προϊόντα μας και σίγουρα μέχρι το 2050 θα χρειαστεί μια αύξηση της παραγωγής 20 έως και 30%. Το θέμα των εισαγωγών μπορεί να είναι πρόβλημα τώρα, αλλά θα πρέπει να εξετάσουμε και τις μελλοντικές εξέλιξεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη γύρανση του γεωργικού πληθυσμού, αυτή είναι γεγονός. Και ακριβώς λόγω της γύρα αυτής, θεωρώ ότι η κοινή οργάνωση αγοράς θα πρέπει να στηρίξει αυτές τις επιχειρήσεις. Γιατί αν οι ε, Γεωργιάνο το 60 ετών ε, πρέπει να σταματήσουν τις γεωργικές δραστηριότητε, έτσι θα απολέσουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, ίσως και το μισό του γεωργικού πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε τις γεωργικές επιχειρήσεις, τους παραγωγούς, για να παραμείνουν στην ε, γεωργική δραστηριότητα. Υπάρχει πρόβλημα με την ηλικία των γεωργών. Αλλά ακόμη και οι πιο ηλικιωμένοι γεωργοί μπορούν κάλλιστα να συνεχίσουν δραστηριότητες και αν τους στηρίξουν οι οργανώσεις παραγόνοι οι συνεταιρισμοί θα ανταποκριθούν πολύ καλύτερα στις απαιτήσεις. Επίσης θα πρέπει να προσελκύσουμε τους νέους ε, στη γεωργία. Γιατί οι νέοι φυσικά προτιμούν σταθερά επαγγέλματα με σταθερό εισόδημα. Κάτι που είναι δύσκολο να έχουμε σταθερό εξασφαλισμένο μηνιαίο εισόδημα στη γεωργία. Επίσης, όταν μιλήσαμε για ασφάλεια, πρέπει να υπάρχει μια εξασφάλιση του εισοδήματος, ιδιαίτερα στους ε, χάλεπους καιρούς. Γι' αυτό είπα τα αμοιβαία κεφάλαια ε, και μια συσπήρωση των γεωργών ώστε να δουν από κοινού, να αποσύρουν προϊόντα σε περίπτωση κρίσεως και να έχουν ένα σύστημα ασφάλισης για να αντιμετωπίζουν τους δύσκολους καιρούς. Έγιναν κάποια τέτοια προγράμματα στην Ιταλία για να εξασφαλιστεί ένα γεωργικό εισόδημα. Υπάρχει ένα πρόβλημα με την εφαρμογή των κανόνων, αλλά ακόμη και κάποιες ασφαλιστικές εταιρείες αρχίζουν και εξετάζουν σοβαρά το θέμα της ασφάλισης της Πρόσφατα είχαμε πρόβλημα στη σχέση και στο σχετισμό δυνάμεων μεταξύ παραγωγής και διάθεση στην αγορά, marketing. Ίσως θα μπορούσαμε να θεσπίσουμε ένα κανόνα θεμητών ή βέλτιστων εμπορικών πρακτικών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ε, εγχειρίδιο στα κράτη-μέλη. Τώρα, σε ό,τι αφορά σχέση παραγωγού, λιανεμπόρου ή αλυσίδα διανομή, είναι σχέση ιδιωτικού δικαίου. Δεν έχει δικαίωμα επέμβαση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά ίσω ένα κώδικα ε, καλών εμπορικών πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο εν μέρει θα μπορούσε να λύσει αυτό το πρόβλημα τη ανισορροπία δυνάμεων μεταξύ παραγωγών και διανομέων. Τώρα, σε ό,τι αφορά την μεταποίηση και τη διαχείριση των κρίσεων ε, και τη δωρεάν διανομή οπωροκυπευτικών προϊόντων, η δωρεάν διανομή ήταν ένα εργαλείο που επινόησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν χρειάζεται να καταργηθεί, αλλά σίγουρα η μεταποίηση είναι επίσης πολύ χρήσιμος μηχανισμός. Και θα βοηθήσει και τους μη οργανωμένους παραγωγούς να χρησιμοποιήσουν κάποιες πηγές χρηματοδότησης. Ε, δύο πράγματα. Η μείωση της κατανάλωσης πρόκειται για τα νοπά οπροκυπευτικά. Αυτόν βλέπουμε τη μείωση στην κατανάλωση. Οι αιτίε είναι πολλαπλές. Καταρχήν ο ανταγωνισμός από τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Ενδεχομένως κάποια ε, ε, δυσκολία στην πρακτική κατανάλωση. Γενικά είναι ακριβά τα προκυπευτικά αν συγκρίνουμε με, ε, θεωρείται ότι είναι ακριβά σε σχέση με άλλα προϊόντα, αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Ε, υπάρχουν όμως αιτίες για τη μείωση. Ο καταναλωτής γνωρίζει τα ωφέλη της μεσογειακής διατροφής, αλλά οι διατροφικές συνήθειες μεταβάλλονται πολύ αργά. Με πολύ αργό ρυθμό. Γι' αυτό χρειάζεται διανομή στα σχολεία, προγράμματα προώθησης, μια συνεχής προσπάθεια για να τροποποιήσουμε σε βάθος τις καταναλωτικές συνήθειες. Δεύτερον, ίσως δεν εκφράστηκα καλά, δεν υποστηρίζουμε την ε, μείωση των δασμών. Ζητούμε απλώς την αμοιβαιότητα. Για παράδειγμα, αμοιβαιότητα με την Τουρκία. Η Τουρκία είναι σημαντικός ε, εξαγωγέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, όταν όμως θέλουμε εμείς να εξάγουμε προκυπευτικά στην Τουρκία, οι δασμοί είναι 50%. Όχι όχι μόνο στην Τουρκία και σε άλλες χώρες. Οπότε ζητούμε την αμοιβαιότητα. Επίσης ε, αμοιβαιότητα και στους ε, όρους για τους εργασιακούς, τους περιβαλλοντικούς και τους άλλες απαιτήσει. Σας ευχαριστούμε. Καταπληκτικές ε, οι παρουσιάσεις, οι μελέτες. Πολύ εύστοχη επιλογή των εμπειρογνωμόνων. Νομίζω ότι πολλά διδαχθήκαμε και θα αξιοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες προς όφελος του κλάδου των απορροκυπευτικών. Ο κύριος Μέλο θα αναλάβει την έκθεση αυτή όπως είπα και ευχαριστούμε θερμά για την οργάνωση αυτού του εργαστηρίου. Και είπαμε ότι στην οργάνωση αγορά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την διαίρεση μεταξύ Βορρά και Νότου και αυτή την περιφερειακή σκόπια, τη σύνθεση του πληθυσμού, την δυνατότητα πιο άμεσης αντίδρασης και επέμβαση σε περίπτωση κρίσης για να αντιμετωπιστούν καλύτερα οι κρίσεις. Γιατί η άμεση δράση είναι το κλειδί ε, της ε, διόρθωσης του προβλήματος. Και η πρόληψη που είναι πολύ σημαντικό γιατί έτσι θα γλιτώσουμε και πολλά έξοδα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ολοκληρώνουμε αυτό το σημείο και περνάμε στο επόμενο. Πολύ σημαντικό και αυτό. Πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε συστηματικές ε, επαφές με εκπροσώπους της Έκσπο. Σήμερα έχουμε την κυρία Λίβια Πομοντόρο, που είναι πρόεδρος του Κέντρου του Μιλάνου για την νομοθεσία και την πολιτική των τροφίμων. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι πέρυσι είχαμε την χαρά να φιλοξενήσουμε τον κύριο Φραντς Φίσλερ, που είναι ο πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής της ΕΞΠΟ του Μιλάνου, και τον καθηγητή Ρικάρτο Βαλεντίνη, πρώην βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, ε, ως μέλος της ε, Διακυβερνητικής Επιτροπής Κλιματικής Αλλαγής. Και σήμερα έχουμε τη χαρά να υποδεχόμαστε την κυρία Λίβια Πομοντόρο, Ο κύριος Δεκάστρο βέβαια εδώ είναι ο πιο αρμόδιος για τα θέματα αυτά. Συστηματικά επαναρχόμαστε στο θέμα της ε, Expo του Μιλάνου για το 2015. Και σήμερα έχουμε μια νέα φάση, ένα νέο στάδιο της ε, συζήτησης για την Expo του Μιλάνου. Είμαστε έτοιμοι και παρακαλώ την κυρία Πρόεδρο του Κέντρου του Μιλάνου να λάβει το λόγο για να μας κάνει την παρουσίαση. Και σας ζητώ ειλικρινά συγγνώμη για την καθυστέρηση που είχαμε στην έναρξη της συζήτησης του δικού σας θέματος. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Και ευχαριστώ για την κατανόησή σας. Προσπάθειά μας είναι να προωθήσουμε την έκθεση αυτή στο Μιλάνο για να δημιουργηθεί και μια συνέχεια συνέχεια μετά την έκθεση του Μιλάνου για τις επόμενες γενναίες. Να προσπαθήσουμε να προωθήσουμε μια πλατφόρμα που θα είναι το πρώτο βήμα για μια πολυμερή διάσκεψη, συγγνώμη, πολυμερή σύμβαση για ε, να υπάρξουν εγγυήσει ότι θα γίνεται σεβαστό το δικαίωμα στη διατροφή. Αυτό το δικαίωμα δεν είναι παντού αναγνωρισμένο και στην πράξη ε, υλοποιείται μόνο σε ορισμένες περιοχές του κόσμου. Φιλοδοξία μας ήταν να καλέσουμε τις Ιταλικές αρχές να παίξουν ηγετικό ρόλο σε μια προσπάθεια να αναγνωριστεί ο ρόλος της έκθεσης. Και αυτό είναι και το σύνθημα της έκθεσης. Για να επιτύχουμε αυτό το στόχο έχουμε βέβαια πολλή δουλειά να κάνουμε. Να συνδέσουμε την έκθεση του Μιλάνου με την έκθεση την αντίστοιχη που θα γίνει στο Ντουμπάι το 2020 και να συμπεριλάβουμε και τους στόχους της χιλιετίας. βασιζόμαστε στην ε, Ιταλική παράδοση. Ε, να μην ξεχνάμε ότι ο Τσέζαρε Μπεκαρία είναι από το Μιλάνο. Πρέπει να αγωνιστούμε λοιπόν για να υπάρχει σωστή διατροφή και να υπάρχει διατροφή στον κόσμο. Έχουμε καναλάβει και άλλες πρωτοβουλίες ε, για την καταπολέμηση του οργανωσμένου εγκλήματος, για να βοηθήσουμε τα άτομα με αναπηρίες, για να αντιμετωπιστεί ο γενετήσιος ακροτηριασμός των γυναικών. Και κατά της θανατικής ε, ποινής έχουμε δραστηριοποιηθεί. Στην Ιταλία είναι επίσης η έδρα και του Παγκόσμιου Οργανισμού Διατροφής. Η Ευρώπη λοιπόν πρέπει να καταλήξει σε έναν κοινό στόχο. Και αυτό επιδιώκουμε σήμερα. Θέλουμε να αποτίσουμε φοροτιμή στην εργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να σας παρακαλέσουμε να υποστηρίξετε τους στόχους που θα μοιραστούμε μαζί σας. Έχουν γίνει πολλές προτάσεις, πολλά ψηφίσματα από το κοινοβούλιο σας που ασχολούνται με το, το θέμα των τροφίμων και της διατροφής και ιδιαίτερα για τα δικαιώματα των ανθρώπων. Για παράδειγμα, στρατηγική για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της ε, διατροφικής αλυσίδας, μέτρα για να μειωθεί η απώλεια τροφίμων ο υποσυτισμός, η ανεπαρκής διατροφή στις αναπτυσσόμενες χώρες, όλα αυτά τα είναι θέματα με τα οποία έχετε ασχοληθεί και που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πιστεύω ότι όλες αυτές ε, οι ιδέες ε, εντάσσονται στα πλαίσια των στόχων της χιλιετίας. στα πλαίσια γενικότερα του πλαισίου για την ανάπτυξη της Ένωσης που ενέκρινε που εγκρίθηκε το 2014 και για την καταπολέμηση της φτώχειας που είναι ο πρώτος στόχος ε, της αναπτυξιακής πολιτικής. Βεβαίω η προσέγγισή μας πρέπει να βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και να εστιάζει στα άτομα. Το θέμα δεν είναι μόνο επιστηστική ασφάλεια η διατροφή είναι ουσιώδες και θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Και όπως ξέρετε, αυτή η τοποθέτηση είναι η τοποθέτηση και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά από πολλές διαβουλεύσεις και υποστηρίζεται πλήρως από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Σε ανακοινώσεις ε, που έχουν εκδοθεί για να εξεταστεί το θεματολόγιο μας μετά το 2015. Πολλά έχουμε ακόμη να κάνουμε και γι' αυτό προέκυψε η ιδέα να υπάρξει αυτό το κέντρο στο Μιλάνο. Ούτως ώστε να συνεχιστεί η εργασία μας για να επιτύχουμε τους στόχους που προανέφερα. Ποιοι είναι λοιπόν, ποιες είναι οι αντιλήψεις μας να βοηθήσουμε αλλαγές μέσω περισσότερης έρευνας για τη σχέση της γεωργίας, ε, των οικονομικών και της διατροφής. Τι θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε να συλλεγεί, να συσσωρευτεί η γνώση με συλλογικό και συνεργατικό τρόπο, με συνεργασία. Να υπάρχει κριτική εξέταση των αποτελεσμάτων της έρευνας που θα βοηθήσει να δούμε κριτικά και τι νομοθεσία υπάρχει στον αυτό, για τα θέματα αυτά. Όλα αυτά με στόχο να γίνουμε σημείο αναφοράς για όσους εργάζονται για τα θέματα αυτά. Ή ουδήποτε είδους εμπειρογνώμονες, ε, επιστήμονες, νομικοί, οικονομολόγοι, πολιτικοί επιστήμονες. Πολλοί ασχολούνται με θέματα που έχουν να κάνουν με τα τρόφιμα και τον επιστημισμό. Άρα θα έχουν μια επιπλέον δυνατότητα μέσω του κέντρου μας και οι κυβερνήσεις για να αντιμετωπίσουν ε, και την ε, τρέχουσα κρίση, η οποία είναι και κρίση επισητισμού. Το κέντρο μας θέλει να παρέχει ε, βοήθεια και τεκμηρίωση όχι μόνο στους νομικούς και άλλους εμπειρογνώμονες, αλλά και γενικότερα. Να υπάρξει δηλαδή περισσότερη συνειδητοποίηση και εντός της κοινή γνώμης. Και η πολιτική και οι άλλοι κοινωνικοί εκπρόσωποι να έχουν τα αναγκαία μέσα για να προσαρμόσουν το κανονιστικό πλαίσιο. Η έκθεσή μας είναι μια θαυμάσια ευκαιρία για να επιτύχουμε αυτό το στόχο. Το Μιλάνο το 2015 είναι η παγκόσμια πρωτεύουσα τροφίμων και διατροφής. Στόχος μας είναι να αναπτύξουμε περαιτέρω αυτή μας την εκδήλωση στρέφοντας τη ματιά μας προς το μέλλον. Ούτως ώστε να διασφαλίσουμε ότι ο στόχος μας να θρέψουμε τον πλανήτη να γίνει στόχος ε, στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης όλων. Να στραφούμε προς το μέλλον σημαίνει να προετοιμαστούμε για το μέλλον. Με βάση την επαγγελματική μου εμπειρία αντιμετώπισα τις δυνάμεις του κακού όπως το διεθνές έγκλημα και άλλους αλλά αντιμετώπισα και τις δυνάμεις του καλού είδα τους εθελοντές που πηγαίνουν στην Αφρική να βοηθήσουν τα παιδιά να προωθήσουν την ανάπτυξη. Η δικαιοσύνη πρέπει να είναι στο κέντρο της προσοχής μας, γιατί είναι τμήμα του πολιτισμού μας αυτή η κουλτούρα της δικαιοσύνης. Στη ζωή μου είχα πολλές δυνατότητες και λόγω των δυνατοτήτων δέχτηκα την ε, πρόταση της ε, έκθεσης του Μιλάνου να κάνω και εγώ την μπορώ τόσο ώστε αυτή η έκθεση Μιλάνου 2015 μην είναι απλώς ε, μια συζήτηση επί των πορισμάτων της έρευνας για τα θέματα αυτά. Αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε είναι να αυξηθεί η συνειδητοποίηση από πλευράς του κοινού ότι πρέπει όλοι να συμβάλλουμε ούτως ώστε ο κόσμος να γίνει καλύτερος. Ε, ξέρω ότι έχω περιορισμένο χρόνο. Συγγνώμη, ενώ ευρύτερα ε, ο χρόνος επήγει για να ε, εφαρμοστούν αυτές οι αλλαγές. Και δύσκολες οι προκλήσεις που έχουμε ενώπιόν μας αλλά θα συνεχίσουμε να εργαζόμεθα σκληρά για να επιτύχουμε τους στόχους μας. Δεν θα αποθαρρυνθούμε από οποιασδήποτε δυσχέρειες. Είμαστε τμήμα της κοινωνίας των πολιτών, θέλουμε ο κόσμος να γίνει καλύτερος. Δεν θέλουμε να τον αφήσουμε χειρότερο ή στο ίδιο επίπεδο με αυτόν που βρήκαμε. Και πώς θα βελτιώσουμε τον κόσμο? Πρέπει να αξιοποιήσουμε το νόμο, να υπάρξει σωστή νομοθεσία, σωστοί κανόνες ούτως ώστε το δικαίωμα στη διατροφή να γίνει ουσιώδες και παγκοσμίως αναγνωρισμένο και εφαρμοζόμενο δικαίωμα. Οπότε, οπότε πιστεύω ότι μπορούμε να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους αν μας στηρίξει συνολικά και η Ευρώπη. Θα κάνουμε τα αρχικά βήματα, αλλά βεβαίως μακρύς είναι ακόμη ο δρόμος ενώπιόν μας για να έχουμε έστω και ελάχιστους κανόνες για τα θέματα αυτά τους οποίους να μπορούν να προσυπογράψουν όλες οι χώρες του κόσμου για να εγγυηθούν τα δικαιώματα όλων των πολιτών στη διατροφή. Βεβαίω μπορεί να φαίνονται μεγαλώστε διακηρύξει, αλλά πολλοί εργάζονται για τον τομέα αυτό. Πολλοί εργάζονται σκληρά, ούτω ώστε να υπάρξει η αναγκαία βάση για να συνεργαστούμε όλοι στην Ευρώπη και στον κόσμο ολόκληρο για να πετύχουμε αυτό το στόχο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Δεκάστρο είναι ο πρώτος μας ομιλητής. Κύριε καθηγητά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όχι μόνο εθιμοτυπικά, κυρία Απομοντόρο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ουσιαστικά και ένθερμα. Να σας ευχαριστήσω επίσης για το έργο του Κέντρου του Μιλάνου. Η Expo Μιλάνου είναι μια μοναδική ευκαιρία, όπως έχουμε πει επανειλημμένως, για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις όλης της ανθρωπότητας, την ε, τροφιμική ασφάλεια και την δυσκολία ανέβρεσης τροφίμων στον κόσμο. Σας άκουσα πολύ προσεκτικά και το έργο σας ε, βρίσκεται μέσα στο ραντάρ μας. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να εγκρίνουμε ένα ψήφισμα, όπως συμφώνησαν χτες οι ε, συντονιστές ε, και η δική σας παρουσία μπορεί να συνεισφέρει. Η Παγκοσμία Έκθεση του Μιλάνου είναι μεγαμοναδική ευκαιρία. Τα θέματα της ε, του Μιλάνου από ε, των δικών μας δραστηριοτήτων. Μιλούμε για, τις, ε, φυσικές, ε, για το φυσικό πλούτο, για το νερό, για τη σπατάλη του, για τη σπατάλη των φυσικών πόρων. Θα ήταν χρήσιμο να εγκριθεί από την Ολομέλεια, από την Ολομέλεια ένα ψήφισμα και για την σπατάλη των τροφίμων. Η Κομισιόν Juncker αντίθετα με την προηγούμενη Επιτροπή Μπαρόσο, έχει, είναι πολύ πιο δραστήρια. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα, τις προκλήσεις του μέλλοντος, το δικαίωμα στην τροφή, η διαχείριση των τροφίμων, η σημαντική αύξηση της παχυσαρκίας ε, στις ανεπτυγμένες ε, και πλούσιες ε, χώρες, ενώ όλα αυτά συνοδεύονται από ε, ύπαρξη ε, ε, φτώχειας και κακής διατροφής για, σε πολλές περιοχές του πλανήτη και στρώματα του πληθυσμού. Η έξπο του Μιλάνου θα μας δώσει την ευκαιρία να ζητήσουμε από τον κόσμο να διαχειριστεί αυτό το παράδοξο. Πρέπει να δράσουμε και σε νομοθετικό επίπεδο. Θα πρέπει να ενοποιήσουμε τους κανόνες ε, στις διάφορες, σε όλες τις ε, ε, υπήρους του πλανήτη, διότι οι διαφορετικοί κανόνες δημιουργούν νομική αβεβαιότητα, δημιουργείται ένας ε, ε, ανταγωνισμός ο οποίος ε, δεν είναι υγιής. Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν κυρία Πομοντόρο. Αν μπορούσατε να μας δώσετε και γραπτό στην παρέμβασή σας θα μας βοηθούσε πολύ. Μάλιστα, ευχαριστούμε. Ο κύριος Τσούλο. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και την Πρόεδρο. Άκουσα... Άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή την παρουσίαση της κυρίας Πομοντόρο και ομολογώ ότι με εξέπληξε θετικά. Γιατί εκτός από τη διασύνδεση που κάνατε με τις ε, επιχειρήσεις, κάνετε προσπάθειες ε, για να αξιοποιήσετε τις ευκαιρίες που δίνει όλη αυτή η οργάνωση της Expo του Μιλάνου για να προωθήσετε ποιοτική διατροφή και υγιεινή διατροφή. Είναι σημαντικά αυτά τα θέματα και συνειφασμένα με τη δημόσια υγεία. Ποιοτική διατροφή, ποιοτικά τρόφιμα σημαίνει ε, και τρόφιμα που πληρούν περιβαλλοντικές, κοινωνικές και ε, προδιαγραφές δεοντολογίας. Όλα αυτά τα θέματα θα ληφθούν υπόψη την έξπο του Μιλάνου για το 2015. Μόνο έτσι θα επιτύχουμε μια πραγματική αλλαγή της νοοτροπίας και της ε, κουλτούρας της διατροφής. Είναι σημαντική λοιπόν η ευκαιρία που μας δίνει η έξπο του Μιλάνου για το 2015 αλλά θα την αξιοποιήσουμε μόνο αν αλλάξουμε τη θεώρηση των πραγμάτων. Γιατί θα πρέπει να προσθέσουμε και μια περιβαλλοντική διάσταση στη διατροφή, κάτι που δεν ίσχυε μέχρι τώρα. Και αυτό πραγματικά θα ήταν ποιοτικό άλμα και προς όφελος της γενικής ε, ευημέρειας. Ελπίζω να μην αμεληθεί αυτό το θέμα στην έξπο του Μιλάνου και να μην περιοριστεί σε μια πανηγυρική εκδήλωση που δεν θα έχει αποτελέσματα μετά το τέλος της διοργάνωσης. Ευχαριστώ κύριος Νταντά. Ευχαριστώ. Θα ήθελα εκ μέρους της ομάδας μου να ευχαριστήσω την κυρία Πομοντόρο για την ομιλία της. Μία διεθνής έκθεση ε, όπως του Μιλάνου του 2015 είναι μία ευκαιρία για να προωθήσουμε την πρόοδο που έχουμε επιτελέσει. Και η Ιταλία με την οικουμενική αυτή έκθεση, την έξπο του Μιλάνου, ε, προτάσει σε κάποια θέματα που μερικοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα θεωρούν παροχημένα. Το θέμα της διατροφής, της ποιότητας της διατροφής, ε, της ε, ε, διαθεσιμότητας των τροφίμων. Είναι πολύ σημαντικά θέματα που θα μας απασχολήσουν και στο μέλλον. Και αναφυσβήτητα θα είναι ένα από τα πιο δυσεπίλητα προβλήματα που θα έχουμε στο μέλλον και πρόκληση εφάμιλη αυτή της ενέργειας. Το γεγονός λοιπόν ότι η Expo του προωθεί αυτά τα θέματα δίνει σημαντικές ευκαιρίες που θα πρέπει να τις αξιοποιήσουμε και στην Επιτροπή μας και να σας στηρίξουμε στις πρωτοβουλίες σας. Γιατί η διατροφή είναι και ένα πολιτιστικό δεδομένο. Και μέσω των εξελίξεων στο Μιλάνο θα στείλουμε ένα χειρό μήνυμα σε ολόκληρη την Ιφίλιο. Και αυτό το μήνυμα θα πρέπει να συνεχιστεί και περαιτέρω και να μην σταματήσει με την ΕΞΠΟ. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για την πρωτοβουλία σας, για την παρουσίαση και σας διαβεβαιώ ότι θα σας υποστηρίξουμε ανεπιφύλακτα στις πρωτοβουλίες αυτές. Σας ευχαριστώ και ως Thank you, Chairman. Uh, I was interested to listen to De Castro, and άκουσα με πολύ ενδιαφέρον τον κύριο Δεκάστρο που μίλησε για τη σπατάλη. Είναι αναφυσβήτητο ότι γίνονται τεράστιες σπατάλες στην αλυσίδα διανομής των τροφίμων και πολλές σπατάλες από τους ίδιους τους καταναλωτές. Τι γνώμη έχετε εσείς για το θέμα αυτό κύριε Πομοντόρο. Η σπατάλη των τροφίμων ε, είναι σημαντικό θέμα φλέγων. Και μάλιστα στο παρελθόν τρέφαμε τα γουρούνια με τα υπολείμματα της διατροφής. Και μάλιστα τα γουρούνια τρέφονταν με τέτοια υπόλοιπα διατροφής, υπόλοιπα τροφίμων και εμεί τρώγαμε τα γουρούνια στη συνέχεια. Καταναλάμε το χοιρινό κρέα. Σήμερα όμω γίνεται λόγο για τη μεταφορά, μόλυνση με ε, διάφορες επιζωτίες. Μάλιστα ο αυθόδης πυρετός ξεκίνησε από, μια, από ένα χειροστάσιο στον Εμένο Βασίλειο. Παρ' όλα αυτά το χοιρινό κρέας είναι θρεπτικό. Ε, πιστεύετε ότι μήπως ε, η σπατάλη των τροφίμων θα λυνόταν με τη χορήγηση των απομιναριών αυτών ε, στα γουρούνια, στα, στα ζώα ή είναι κάτι που ανήκει στο παρελθόν και δεν πρόκειται να εφαρμόσουμε μια τέτοια μέθοδο. Επίσης, ε, στα σφαγεία γίνονται φοβερές σπατάλες και τα υπολείμματα των σφαγείων, ακριβώς επειδή είχαν πολλές πρωτεΐνες, εντάσσονταν στις, ενσωματώνοντας τις ζωοτροφές. Τώρα όμως σε καμία περίπτωση λέμε ότι θα πρέπει να τρέφουμε ζώα με ε, υπολείμματα ζωικά του ίδιου ζωικού είδους. Για, παράδειγμα στα μυρικαστικά. Γιατί όμως να μην δίνουμε προ, πρωτεΐνη μυρικαστικό σε πουλερικά ή χοιρινά και ε, το ανάπαλιν. Από τη στιγμή που γίνεται διασταύρωση, μάλλον περνάμε το ζωικό είδος, δεν έχουμε την προϋπόθεση αυτή ότι δεν πρέπει να τρέφουμε ζώα με συγγενικά του ζώα. Τι γνώμη έχετε γι' αυτό. Γιατί έχουμε σπατάλη, έχουμε τέτοια απόβλητα, τέτοια απομεινάρια και υπάρχει δυνατότητα διοχέτευσή του. Γιατί να μην τα αξιοποιήσουμε. Ναι, αλλά αυτά τα τρόφιμα δεν ήταν ομάτα, μαγειρεύαμε. Οπότε του δίναμε μια νέα αξία και μια νέα ποιότητα. Δεν ήταν απλώ υπολείμματα ασφαγείων. Γινόταν μια μεταποίηση, μια θερμική επεξεργασία. Αυτά μας διδάσκει η ιστορία. Η κυρία Πάουλσεν. Ευχαριστώ πολύ και καλωσορίζω την ε, προσκεκλημένη μας. Λοιπόν, το μέλλον της ανθρωπότητας επειδή είμαστε 7,5 δις στον πλανήτη και σε 20-30 χρόνια θα είμαστε ίσως 10 ή 11 δις. Οπότε, επειδή μόνο ένα πλανήτη έχουμε και δεν θα μεγαλώσει και δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να πάμε σε άλλον. Άρα, είναι τρομερή πρόκληση αυτό που αντιμετωπίζουμε. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή, Πρέπει να έχουμε παρκές νερό, πόσιμο νερό. Πρέπει να έχουμε ψάρια στις θάλασσές μας, να διατηρήσουμε τη βιοπικιλότητα. Και επίσης πρέπει να παράγουμε αρκετά τρόφιμα για όλους. Άρα πρέπει να είναι πολύ πιο αποτελεσματική η παραγωγή τροφίμων από ό,τι σήμερα. Ένα το κρατούμε. Αλλά ξέρετε, εγώ θυμάμαι ακόμη το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Γιατί ήμουν παιδί τότε και πεινούσα. Άρα με συγκινεί ιδιαίτερα αυτό που προσπαθείτε να επιτύχετε, αυτό που είπατε αυτό που συζητάμε για την αλληλεγγύη, για την ποιότητα. Φυσικά πρέπει να προστατεύουμε και την ποιότητα. Αλλά, αλλά, υπάρχουν πολλοί παχύσαρκοι. Ενώ τα μικρά παιδιά στον κόσμο πεθαίνουν από την πείνα. και όχι και πολύ μακριά. Αν πάτε στα στρατόπεδα προσφύγων στο Λίβανο θα δείτε ότι δεν υπάρχει η διατροφή που χορηγείται στους πρόσφυγες. Βασίζομαι λοιπόν ε, στις δικές μου εμπειρίες. Θυμάμαι ότι ήμουν παιδάκι πέντε ετών και πεινούσα πολύ και όταν ε, επανήλθε η ειρήνη τότε θεωρούσα α, τώρα θα έχω αρκετό φαΐ. και αν ε, ε, φάω πολύ θα γίνω όμορφη θεωρούσα να πάχαινα. Σας ευχαριστώ πολύ συγκινητικά αυτά που μας είπατε. Ο κύριος Ροπέ είναι ο τελευταίος μας ομιλητής. Ε, ačiū pirmininkė, iš tikrųjų manau, kad labai įdomus ir vertingas. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση της κυρίας Πομοντόρο. Το δικαίωμα στην τροφή είναι πολύ σημαντικό. Καμιά φορά μιλάμε και για το δικαίωμα στο πόσιμο είδωρ και αυτό αποτελεί ε, απαραίτητο κομμάτι της διατροφής. Θα ήθελα να θα σας ρωτήσω αν έχετε και κάποιες προτάσεις. Γιατί ε, υπάρχουν αντικρώμενες, ε, μάλλον υπάρχουν μεγάλες διαφορές ε, στο μέσο εισόδημα, στην ποιότητα ζωής ανάμεσα στην Ευρώπη και άλλες περιοχές του κόσμου. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να φάνε ό,τι θέλουν κάθε μέρα, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι ζουν κάτω από το κατόφλι της φτώχειας. Οπότε χρειάζονται άλλες πολιτικές προφανώς. Πώς πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε να ε, διασφαλίσουμε το δικαίωμα στην σωστή διατροφή, την επαρκή διατροφή, ε, με βάση ένα συγκεκριμένο ελάχιστο αριθμό θερμίδων ε, που χρειάζονται οι άνθρωποι για να ζήσουν με βάση τα ελάχιστα μερομίστια στην Ευρώπη. Έχουμε ανθρώπους με αναπηρία έχουμε ανθρώπους που ζουν μόνοι τους χωρίς οικογένειες να τους βοηθήσουν. Πώς πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε να ε, το εξασφαλίσουμε το δικαίωμα στην πράξη έτσι ώστε να μην είναι μόνο ευχολόγια αυτά που λέμε. Ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε το γύρο των ομιλητών. Παρακαλούμε την καλεσμένη μας αν θέλει να σχολιάσει αυτά που άκουσε. Έχει το λόγο. Χαίρομαι που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία, Πρόεδρε. Οι ερωτήσεις που μου υποβλήθηκαν δείχνουν ότι πρέπει να προετοιμαστούμε καλά. Η ευκαιρία της ε, Expo 2015 δεν συνίσταται μόνο στο θέμα της έκθεσης, αλλά και στο γεγονός ότι είναι ευκαιρία να κάνουμε τη σύνδεση ε, με διάφορα προβλήματα που αφορούν την φύση, το περιβάλλον, το νερό, τα μέσα παραγωγής ε, και τη διανομή της τροφής. και η βιοπικιλότητα ακόμα είναι πρόβλημα. Υπάρχουν χώρες ε, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που παράγουν με πολύ μεγάλη απόδοση και κερδοφορία αλλά που προκαλούν σημαντικά, σημαντικές ζημίες στο περιβάλλον. Έχω σπουδάσει δραματική και γνωρίζω πολύ καλά πώς μπορούμε ε, να, και πώς μπορεί η ίδια έκθεση του Μιλάνου να γίνει ε, να παρουσιαστεί ως ένα δράμα εντυπωσιακό ε, και συγκινητικό αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να έχει και ένα νόημα για όλη την ανθρωπότητα γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε όλα να μείνουν στη βιτρίνα. Πρέπει λοιπόν να υποφεληθούμε από την ευκαιρία. Γι' αυτό το λόγο βρίσκομαι εδώ σήμερα μαζί σας. Με συγκινεί η αλληλεγγύη σας. πρέπει να αλλάξουμε την εστίαση μας. Πολιστικά μιλώ ε, από πολιτικής πλευράς, την εστίαση μας στα προβλήματα της ανθρωπότητας. Υπάρχουν δυσκολίες ακόμα και στην επιβίωση μεγάλων τιμάτων του πληθυσμού. Και μετά έχουμε και πιο ειδικά προβλήματα για ε, τα οποία δεν με ρωτήσατε σήμερα, αλλά θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε τη σύγχυση ανάμεσα στην, ε, στις διακηρύξεις και στην πρακτική δουλειά. Γιατί καλές διακηρύξεις, αλλά θα πρέπει να δουλέψουμε κιόλας για να παράγουμε αποτέλεσμα. Ιδιαίτερα όταν μιλάμε για το δικαίωμα στην τροφή, Ας έχουμε στο μυαλό μας ότι ο πλανήτης μας είναι ενιαίος, είναι ο ίδιος για όλους. Τον καταστρέφουμε σιγά σιγά αυτή τη στιγμή, καταστρέφουμε τη φύση, την κακομεταχειριζόμαστε και σφετεριζόμαστε τους πόρους της Οπότε, τι θα κάνει η ανθρωπότητα μπροστά σε όλα αυτά τα προβλήματα και στο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. Τι θα κάνει ε, ενώπιον του προβλήματος της βιοπικιλότητας. τι θα κάνει με τις αυξανόμενες ανάγκες ε, ε, διατροφής ε, σε ένα κόσμο του οποίου οι φυσικοί πόροι μειώνονται. Πρέπει να το συζητήσουμε και να συμφωνήσουμε μεταξύ μας. Το... Στην αρχή είχαμε όνειρα και εγώ είμαι αισιόδοξο άτομο αλλά δεν αρκούν τα όνειρα. Πρέπει να σηκώσουμε τα μανίκια για να δουλέψουμε. Και γι' αυτό χρειάζεται ουσιαστική αλληλεγγύη. Χρειαζόμαστε ε, προγράμματα για να εγκαθιδρύσουμε ελάχιστους κανόνες, όπως τους ονομάζει ο ΙΕ, ε, που θα την χάνουν σεβασμού σε όλο τον κόσμο. Γιατί αν έχουμε ελάχιστες προδιαγραφές, ε, οι οποίες ακολουθούνται εδώ και όχι εκεί, ε, θα έχουμε αποτύχει. Μετά χρειάζεται να διαθέτουμε πραγματικά θεμελιώδη δικαιώματα, τα οποία να τη χάνουν σεβασμού παντού, σε όλο τον κόσμο. Ο δρόμος είναι μακρύς, το ξέρω. Και γνωρίζουμε και τα όρια μας. Ξέρουμε μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε. Αλλά πάντως θα πρέπει να δείξουμε αλληλεγγύη. Θα πρέπει να δώσουμε, να τονίσουμε την ανάγκη να διαθέτουμε ελάχιστες προδιαφές, ελάχιστους κοινούς κανόνες για όλο τον κόσμο. Ένα παράδειγμα σας δώσω. Το 2020 το Ντουμπάι θα φιλοξενήσει την έξπο, την έκθεση των τεχνολογιών της καινοτομίας. Δεν θα μπορούσαμε ήδη να δημιουργήσουμε μια γέφυρα ε, με την Expo 2020. Γιατί η καινοτομία θα μπορούσε να μας βοηθήσει να λύσουμε ορισμένα πρακτικά θέματα. Μιλήσαμε για την σπατάλη των τροφίμων και το πώς θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ε, απόβλητα, ε, υπερισεύματα, οζοτροφή στο Σικάγο πριν από κανένα αιώνα. Συνεδρίασε το 1893 με την ευκαιρία της ε, έκθεσης του Σικάγου, της έξπο του Σικάγου, ε, υπήρχαν ε, εκτάσεις ε, οι οποίες ήταν ε, βρώμικες, βρωμούσαν πραγματικά και εκεί χτίστηκε ε, το μεγάλο κέντρο το οποίο φιλοξένησε την ΕΞΠΟ. τα υπολείμματα των σφαγίων χρησιμοποιήθηκαν όχι μόνο για ε, ζωοτροφές μυρικαστικών αλλά και για λιπάσματα. Λιπάσματα τα οποία οδήγησαν στη δημιουργία πολύ πλούτου. Λάθος επιλογή. Δεν μπορώ να πω πολλά γι' αυτό, αλλά το πρόβλημα των υπολοιμάτων ε, τροφής ε, όπως επίσης και το πρόβλημα το ότι κάποιοι έχουν πάρα πολύ τροφή και κάποιοι καθόλου, ε, μας ε, φέρνει στη συζήτηση αυτή που έχει δύο όψεις και θα γίνει και στο Μιλάνο. Πώς θα πολεμήσουμε, πώς θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της σπατάλης τροφών ε, ή της δημιουργίας, να το δούμε αλλιώς, του ελάχιστου, της ποσότητας αποβλήτων και από την άλλη μεριά του πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα απόβλητα για να παράγουμε κάτι πιο χρήσιμο. Δεν είναι το δικό μου θέμα, δεν, είμαι, δεν συνηθίζω να δίνω συμβουλές για πράγματα που δεν γνωρίζω σε βάθος, οπότε δεν θα πω τίποτα γι' αυτό, αλλά το πρόβλημα, τα προβλήματα αυτά που είναι έτσι γενικά όπως η σπατάλη των τροφίμων και το πρόβλημα των αποβλήτων θα πρέπει να, να αντιμετωπίζονται και θα το κάνουμε, θα το συζητήσουμε στην πλατφόρμα της Expo του Μιλάνου. Τελειώνω Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Θα ζητώ συγγνώμη αν σας καθυστέρησα. Να προσθέσω μόνο ε, μία ακόμα φρασούλα. Η ε, νιώθουμε, έχουμε, ε, η πορεία προς την έξοδο του Μιλάνου ήταν τόσο μακρά που νιώθουμε σαν να έχει ήδη γίνει. Ε, η πορεία αυτή χρειαζόταν γνώση, χρειαζόταν έρευνα, χρειαζόταν πολλή δουλειά, χρειάστηκε και ε, συνεργατική προσπάθεια. Ε, χρειάστηκε να συνδυάσουμε τη γνώση τόσων πολλών ανθρώπων με τις ανάγκες όλης της ανθρωπότητας. Ε, θέλουμε να αποφύγουμε ε, την καταλήστευση των ε, πόρων, των φυσικών πόρων προς όφελος μόνο ελάχιστον. Θα ήθελα τελειώντας να σας ζητήσω να μας βοηθήσετε και ως Επιτροπή Γεωργίας αλλά και γενικότερα ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλουμε να συνδυάσουμε τις γνώσεις, τις εμπειρίες όλων και να ζητήσουμε λύσεις που θα δώσουν αποτελέσματα για όλους και όχι μόνο για λίγους. Σας ευχαριστούμε θερμότατα, κυρία Παμοντόρο. Πολύ καλό το μήνυμα και πολύ εύστοχη η ανακεφαλαίωση του κυρίου Νταντά που είπε ότι από το Μιλάνο θα εκπορευθεί ένα μήνυμα προς ολόκληρη την Ιφίλιο. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Μιλήσαμε για το περιβάλλον, για την ενέργεια, για την καινοτομία, την διάδοση της γνώσης. Όλα αυτά λαμβάνονται υπόψη στο κέντρο του Μιλάνου, στο οποίο προεδρεύεται και Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό. Ο κύριος Δεκάστρο είναι ο δικός μας ε, πρέσβης και αντιπρόσωπος στην έξπο του Μιλάνου, οπότε θα μας ενημερώνει τακτικά για τις πρωτοβουλίες και τις εκδηλώσεις εκεί, προκειμένου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρακολουθεί και να ε, συμμετέχει ενεργά για τη, στη διαμόρφωση αυτού του σημαντικού μηνύματος που θα πρέπει να στελεί από την έξπο του Μιλάνου σε ολόκληρο τον κόσμο. Ολοκληρώσαμε το σημείο αυτό και περνάμε στο επόμενο. Το σημείο 14 που προβλέπει μια σύντομη παρουσίαση από τη Γενική Διεύθυνση της Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικής Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες που διαθέτει εν λόγω Γενική Διεύθυνση για τη στήριξη της εργασίας των Επιτροπών. Η νέα Γενική Διεύθυνση ε, συστήθηκε την 1η Νοεμβρίου του 2013. Η Γενική αυτή Διεύθυνση συνένωσε ε, ήδη προϋπάρχουσες ε, υπηρεσίες και διευθύνσεις που στόχο είχαν τη στήριξη των, Ευρωβουλευτών ή των Επιτροπών. Είχαμε τη Γενική Διεύθυνση της, τη διεύθυνση, συγγνώμη, της Βιβλιοθήκης, την πρώην Γενική Διεύθυνση Πρέσ την Διεύθυνση για την Ανάλυση των Επιπτώσεων και της Προστιθέμενης Αξίας, πρώην Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών και προσθέθηκε και μια τελείως νέα διεύθυνση, το, το Γραφείο Αναλύσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ε, προσφέρει εξατομικευμένη ενημέρωση και έρευνα στους ευρωβουλευτές και μια σειρά συνοπτικών δημοσιευμάτων προς τους ευρωβουλευτές. Επίσης ε, γίνονται αναλύσεις ε, και χορηγούνται αμερόληπτες και ανεξάρτητες ε, έρευνες ε, και τα πορίσματά προς τους βουλευτές για την άσκηση της κοινοβουλευτικής τους δραστηριότητας. Είναι ικανότητες εφάμιλες αυτές που προσφέρονται και σε άλλες κοινοβουλευτικές δημοκρατίες. Οπότε είναι σημαντική αυτή η Γενική Διεύθυνση για τον εξάντα και εξπόστ ε, έλεγχο και την ε, μελέτη επιπτώσεων, ε, για την ευρωπαϊκή προσθεμένη αξία, την επιστημονική επισκόπηση, την γενική, τον γενικό έλεγχο και την εποπτεία του Συμβουλίου και την εκτίμηση των επιδόσεων. Έχουμε τον κύριο Γιώζεφ Ντούν που προσφέρθηκε να έρθει στην Επιτροπή και να μας παρουσιάσει μερικές δραστηριότητες αυτής της νέας Γενικής Διεύθυνσης. Ο κύριος είναι ο, ο Σκον, τα καθήκοντα διευθυντού στην EPRC. Αν δεν προλάβετε να δώσετε όλα τα στοιχεία στην προφορική σας παρατήρηση, ελπίζω να στείλετε και γραπτός την παρουσίασή σας. Παρακαλώ, κύριε. Ευχαριστώ. Εκπροσωπώ την μία γενική διεύθυνση που δημιουργήθηκε πριν από λίγο πάνω από ένα χρόνο. Όπως είπατε, έχει τρία τμήματα η βιβλιοθήκη που προϋπήρχε. Μία εντελώ νέα υπηρεσία που λέγεται Υπηρεσία Ερευνών για τα μέλη που θέλει να κάνει ενημερώσεις ε, με την τελευταία λέξη των γνώσεων για τα θέματα για τα μέλη και το τρίτο τμήμα είναι για μελέτες επιπτώσεων και ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Στόχος της Γενικής Διεύθυνσης γενικά είναι να βοηθάει τις επιτροπές στην προσπάθειά τους ε, να ελέγχουν και να επιβλέπουν και να δίνει μια τεκμηρίωση για τη δουλειά του. Αυτή λοιπόν η Γενική Διεύθυνση δημιουργήθηκε με βάση την επιχειρηματολογία ότι το Κοινοβούλιο είναι πολύ καλό από πλευράς νομοθετικής υποβολής τροπολογιών αλλά ίσως όχι τόσο ισχυρό στην προπαρασκευαστική ή μετέπειτα φάση. Θέλουμε λοιπόν να ε, προωθήσουμε μια πολιτική κύκλου, μια προσέγγιση κύκλου πολιτικής για την ε, δουλειά του Κοινοβουλίου. Πώς θα βοηθήσουμε λοιπόν την Επιτροπή σας όπως όλες. Πρώτον, κοιτάζοντας μπροστά, δηλαδή μια δουλειά διερεύνησης του τι μπορεί να κάνουμε στο μέλλον. Έχουμε κάποιε εκθέσει πρωτοβουλία που λέγονται Ευρωπαϊκέ Αποτιμήσει που βασίζονται στο άρθρο 225 τη συνθήκη που δίνουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έμεσα τη δυνατότητα πρωτοβουλία. Χωρί να αφαιρούν ε, το δικαίωμα πρωτοβουλία ε, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριο Δεκάστρο είπε στην προηγούμενη συζήτηση ότι περίμενε ο κύριο Γιούγκερ να κάνει προτάσει για ένα θέμα τροφίμων. Αν δεν υπάρξουν τέτοιες προτάσεις από την Κομισιόν, τότε θα μπορούσαμε εμείς να επιδιώξουμε δικαίωμα πρωτοβουλία με βάση το άρθρο 25 για να πιέσουμε την Κομισιόν να υποβάλει και εκείνη προτάσεις. Προτάσεις που να βασίζονται στις απόψεις της Επιτροπής σας. Δεύτερον, για να προβλέψουμε το μέλλον, έχουμε μία αποστολή να βοηθήσουμε τις Επιτροπές να κάνουν ποσοτικές εκτιμήσεις για το τι σημαίνουν οι προτεραιότητές τους. Κάνουμε χθε λοιπόν για το κόστος της μη Ευρώπης για παράδειγμα, για ένα τομέα ή γενικότερα. Στον τομέα της άμυνας για παράδειγμα, αν δεν έχουμε πλήρη ενιαία αγορά, προσπαθούμε να ποσοτικοποιήσουμε τι κοστίζει αυτό με βάση το πνεύμα της παλιάς έκθεσης τσεκίνη του 88. Και κατόπιν έχουμε και το ΣΤΟΑ που επίσης κάνει δουλειά μέλλοντος. Και χαίρομαι που είναι εδώ η κυρία Πέτερ η οποία είναι ενεργό μέλος του ΣΤΟΑ. Το ΣΤΟΑ σας υπέβαλε πέρυσι μια έκθεση για τις ε, τεχνολογικές προκλήσεις της διατροφής 10 δις ανθρωπίνων όντων. και με βάση αυτά που είπε και η κυρία Πομοντόρο ίσως θα σας ενδιέφερε να εξετάσετε περισσότερο τον τομέα αυτό με βάση τις δυνατότητες που σας παρέχει το ΣΤΟΑ. Άλλος τομέας εργασίας επιπτώσεις, ε, μελέτες επιπτώσεων ex post για την εφαρμογή κάποιων μέτρων. Για παράδειγμα, πέρυσι το φθινόπωρο κάναμε μία σύντομη αποτίμηση της εφαρμογής για τα βιολογικά προϊόντα και την σήμανσή τους. Εδώ είναι μία αρχική λοιπόν αποτίμηση. Τα αποκαλούμε αρχικές αποτιμήσεις. Είναι, βασίζονται στις μελέτες επιπτώσεων της Κομισιόν, προσπαθώντας ε, να διαπιστώσουμε που μπορεί να υπάρχουν αδυναμίες. Για την εφαρμογή λοιπόν της νομοθεσίας και των μέτρων, πέρα από αυτές τις εκτιμήσεις εφαρμογής, θέλουμε να στηρίξουμε τις εκθέσεις όταν κάνετε εκθέσεις εφαρμογής. Ξέρετε ότι είναι εκθέσεις πρωτοβουλίας, άρα δεν υπόκεινται σε ποσοστώσεις. Παλιά μπορούσαν να κάνουν επιτροπές μόνο μία τέτοια έκθεση το χρόνο αλλά τώρα έχουν καταργηθεί αυτοί οι περιορισμοί από τη διάσκεψη των Πρόεδρων Επιτροπών και μετά τη διάσκεψη των Πρόεδρων. Είναι λοιπόν μια δυνατότητα που έχετε στη διάθεσή σας για να μπορέσετε να εκτιμήσετε τι έχει συμβεί και μπορούμε να σας υποβάλουμε εκθέσεις ε, τεκμηριωμένες. Βεβαίως, ε, εάν καταλάβουμε καλύτερα πώς εφαρμόζονται οι νόμοι μας, κατόπιν θα προτείνουμε και θα εγκρίνουμε και καλύτερους νόμους στο μέλλον. Και τέλος, τρίτος τομέας, εξάντε μελέτες επιπτώσεων, μελέτες αντικτύπου, για να στηρίξουμε τις επιτροπές. Στην πρώτη φάση εξέτασης, ε, όταν λαμβάνετε τη μελέτη επιπτώσεων, τη μελέτη αντικτύπου, της Κομισιόν σας κάνουμε μία ανάλυση και βοηθάμε τις επιτροπές σας με πιο λεπτομεριακές μελέτες αντικτύπου εάν η επιτροπή σας θεωρεί ότι χρειάζεται επιπλέον δουλειά περισσότερη λεπτομέρεια ότι κάποιος τομέας δεν έχει καλυφθεί από τις ε, μελέτες αντικτύπου της Κομισιόν. Και Κάνουμε και μελέτες αντικτύπου επιτροπολογιών, όχι πολύ συχνά, αλλά λαμβάνουμε όλο και περισσότερα αιτήματα από επιτροπές για τέτοιες ε, μελέτες αντικτύπου σημαντικών επιπτω... ε, τροπολογιών. Βεβαίω είναι σημαντικό αυτό γιατί αν οι τροπολογίε σας ας πούμε φτάσουν στον τριμερή διάλογο τότε αν έχετε και μια αιτιολόγηση των επιπτώσεών τους μπορεί να σας βοηθήσει στις διαπραγματεύσεις και βοηθάει και στη διαφάνεια. Είναι καλύτερη αιτιολόγηση τροπολογιών που αποκλίνουν ριζικά από τις προτάσεις της Κομισιόν. Αυτές βέβαια τις ε, δίνουμε σε εξωτερικούς φορείς γιατί αυτός είναι ο κανόνας που ε, ενέκρινε η διάσκεψη των Προέδρων για λόγους ανεξαρτησίας Μπορούμε να σας βοηθήσουμε λοιπόν με την εφαρμογή, με τη μελέτη της εφαρμογής νομοθεσίας. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε με νομοθετικές εκθέσεις πρωτοβουλίας. Θέλουμε να σας δίνουμε τακτικά βοήθεια για όλα τα θέματα των μελετών αντικτύπου. Έχουμε συνεργαστεί με πολλές επιτροπές μέχρι στιγμής και τη δική σας. Και έχουμε εδώ μία επιλογή έξω των ε, μελετών που έχουμε εκπονήσει θα δείτε ότι ορισμένες είναι πολύ τεκμηριωμένες. Συνοψίζουμε εκεί εργασίες τεσσάρων πέντε φορέων και νομίζουμε ότι είναι και πολύ συγκεκριμένες αυτές οι μελέτες και βοηθούν την εργασία σας. Ελπίζω να ήμουν αρκετά αναλυτικός αλλά να μην μακρηγόρησα και στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και ευχαριστούμε και για το υλικό που μας παρέχετε. Και το χρησιμοποιώ πραγματικά γιατί έχει μεγάλη αξία και επιστημονική και τεχνική. Σας ευχαριστούμε θερμά λοιπόν για αυτή σας την προσφορά. Ο κύριος Ροπέ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τις χρήσιμες πληροφορίες που μας δώσατε. Είναι πραγματικά πολύ ωφέλιμη αυτή η υπηρεσία έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα απονήματα της είναι ιδιαίτερα αξιόλογα. Είναι ευρύτατο το φάσμα δραστηριοτήτων αυτή της υπηρεσία. Στην πράξη όμω τι γίνεται. Ποιο απευθύνεται σε εσά, ε, οι βουλευτές απευθεία ή μια κοινοβουλευτική επιτροπή. Μπορούμε ε, να επικεντρωνόμαστε στις συγκεκριμένες πτυχές του προβλήματος ή θα πρέπει να σας θέτουμε ερώτηση για το σύνολο του προβλήματος και κάνετε και εξωτερική ανάθεση μελετών. Πόσο στοιχίζουν όλα αυτά και πώς τα οργανώνετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Διευθυντά. Θα είχατε την καλοσύνη να απαντήσετε. Μάλιστα. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Μελέτης Επιπτώσεων και της Ευρωπαϊκής Προσθέμενη Αξίας ε, εξυπηρετεί μόνο επιτροπές όχι με μονομένους βουλευτές, γίνεται με τα απαίτημα συγκεκριμένων επιτροπών και συνήθως οι συντονιστές οι επιτροπές αποφασίζουν να ζητήσουν μελέτη επιπτώσεων ή μελέτη επιπτώσεων συγκεκριμένων τροπολογιών. Το αίτημα γίνεται, υποβάλλεται από κοινοβουλευτικές επιτροπές. Τώρα, για νομοθετική ή έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας, αυτόματα η υπηρεσία μας σας προετοιμάζει ε, μία μελέτη επιπτώσεων και προστιθέμενης αξίας και μάλιστα προσαρμόζουμε το περιεχόμενό μας ε, στις συγκεκριμένες πτυχές ε, της έκθεσης και της Επιτροπής. Και εστιαζόμαστε σε επιχειρήματα που σας χρησιμεύουν. Επίσης, ε, το... η Υπηρεσία Κοινοβουλευτικής Έρευνας έχει περισσότερες περισσότερους πόρους και ανταποκρίνεται σε εξατομικευμένες δηλώσεις ε, συγκεκριμένων βουλευτών. Αυτό είναι, αυτή είναι άλλη διεύθυνση της γενικής, γενικότερης διεύθυνσης. Πάντως, περιορισμοί δεν υπάρχουν στο εύρος των ετοιμάτων. Υπάρχει όμως διαφορά μεταξύ αιτήματος ενημέρωσης και συγκεκριμένης ε, αναφοράς ε, ο προπολογισμό μα ετησίων είναι κάτω από ένα εκατομμύριο ευρώ, γύρω στου 900.000 και μάλιστα για όλε τι επιτροπέ. Γενικό προπολογισμό δεν είναι αρκετά δαψίλη όσο ε, φαίνεται ίσω εκ πρώτη όψεω. Ε, όλα εξαρτώνται από τον αριθμό των ετοιμάτων που λαμβάνουμε. Ελπίζω να απάντησα στην απορία σας. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι και οι υπηρεσίε της βιβλιοθήκης ε, έχουν εξελιχθεί ιδιαίτερως και το υλικό που παρέχει η βιβλιοθήκη είναι πολύ πιο ευανάγνωστο, πολύ πιο εύχριστο και παρακαλώ διαβιβάστε <clears throat> αυτά τα συγχαρητήρια και τα κομπλιμέντα στους αρμοδίους της βιβλιοθήκης γιατί πραγματικά έχει αναβαθμιστεί η προσφορά των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης. Και επειδή βρισκόμαστε στην αρχή τη κοινοβουλευτική θητεία, είναι σημαντικό να έχουμε όλε αυτέ τι πληροφορίε που μπορούμε να τι αξιοποιήσουμε στην κοινοβουλευτική μα εργασία, στο κοινοβουλευτικό μα έργο. Γιατί οι δυνατότητε είναι απεριόριστε πραγματικά. Οπότε καλό θα ήταν να, να ετοιμάσουμε ένα έγγραφο με όλες αυτές τις πληροφορίες και να το μοιράσουμε στου ευρωβουλευτέ για να μάθουν τι δυνατότητες έχουν. Γιατί σήμερα είναι πέμπτη τελευταία μέρα της συνεδρίασης που ήταν πολύ έντονη τις προηγούμενες μέρες. Γι' αυτό δεν έχουμε αθρώα προσέλευση ευρωβουλευτών, αλλά θα είναι πολύ χρήσιμο το έγγραφο με τις σχετικές πληροφορίες που θα το προωθήσουμε. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο. Α, συγγνώμη, η κυρία Πετήρ. Κυρία Πετήρ, σύντομα θα ήθελα ως ε, εκπρόσωπος της Άγκρης της ΣΤΟΑ να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μου κάνατε και να επενέσω τις υπηρεσίες αυτές και να σας πω ότι είμαι στη διάθεσή για περαιτέρω συνεργασία για ό,τι κρίνει η Επιτροπή Γεωργίας ότι θα πρέπει να προωθήσουμε στο πάρελ της ΣΤΟΑ και επίση ε, θα ήθελα να μου κάνετε και προτάσει για συγκεκριμένα θέματα που θα θέλατε να προτείνω στη ΣΤΟΑ για να εξεταστούν. Ευχαριστώ. Ε, Σας ευχαριστούμε κύριε Πετήρ. Πραγματικά η συνεδρίασή μας ήταν πολύ πλούσια αυτή τη φορά. Έβριθε θεμάτων σημαντικών και ίσως θα πρέπει να δούμε και τι θέματα θα προτείνουμε για μελέτες. Ανάλογα με τις ε, προσδοκίες μας ε, για το μέλλον της κοινή γεωρικής πολιτικής, ε, ιδιαίτερα μέχρι το 2020. Οι συντονιστές κατέληξαν σε συστάσεις στη χθεσινή του συνεδρίαση τις λάβατε και γραπτός και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Κοιτάξτε αν έχετε παρατηρήσεις, ε, ε, καλώς. Αλλιώς θα θεωρηθούν συγκεκριμένες οι συστάσεις των συντονιστών. Τώρα, επόμενες συνεδριάσεις. Στις 27 Ιανουαρίου, όπως ξέρετε, 3 με έχουμε την έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής με μια δημόσια ακρόαση για το πακέτο του γάλακτος και τις προοπτικές του γαλακτοκομικού τομέα. Ιδιαίτερα σημαντικό και δύσκολο θέμα. Ε, σίγουρα θα είναι και πλούσια μερή σε διάταξη και θα ταλανιστούμε και θα έχουμε μόνο μονόλεπτες ε, ε, παρεμβάσεις και οι τακτικές μας συνεδρίες 23 και 24 Φεβρουαρίου, 3 με 6,5 και 9 με 12.30 και 3 με 6.30. Αν δεν έχετε άλλα σχόλια, κυρίσω το πέρας της συνεδρίασης. Ε, μας περίσεψε και λίγος χρόνος. Δεν χρειάστηκε σήμερα να είμαι πολύ αυστηρός και να κόβω το λόγο μερικές φορές όπως έγινε χθε. Ξέρω ότι αυτό δυσαρεστεί πολλούς, αλλά τι να κάνουμε, αυτό είναι το άχαρο έργο του Προέδρου μερικές φορές. Σας ευχαριστώ, καλή επάνωδο στις πατρίδες σας, καλό ταξίδι και ραντεβού στην επόμενη μας έκτακτη συνεδρίαση με τη δημόσια κρόση για το γάλα. Σας ευχαριστώ όλους και τους διερμηνείς και τους καλεσμένους και τους ευρωβουλευτές και καλή σας όρεξη.